Let's uh, Ας αρχίσουμε γιατί είναι πολύ φορτωμένο το πρόβλημα. Περιμένουμε σιγά σιγά να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους σας. Θα... Σας έχει διανεμηθεί η, η ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις Μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνεται. Στο σημείο 14, εμπόριο και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, αιτήση του κυρίου Μετίν Καζάκ θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα στη θέση του σημείου 12 και το 12 θα πάρει τη θέση του 14. Απλώς έχει αλλάξει η σειρά τους, λοιπόν, 12 με 14. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι και πάλι αναμεταδίδεται το ίντερνετ η συνεδριασή μας Θα έχουμε και μια έκτακτη συνάντηση στο Στρασβούργο με μέλη της Επιτροπής που συμμετείχαν στην ε, συνεδρίαση στην, στην Επιτροπή η οποία έχει γίνει για την ε, ε, έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Έχει αλλάξει η αρχική ημερομηνία. Ούτως ή άλλως έχετε τις σχετικές επεξηγηματικές επιστολές στους φακέλους σας. Και αν έχετε κάποιο θέμα να θέσετε μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε εδώ τον Μάικλ Τόπινγκ μέλος της γραμματείας μας ο οποίος θα πάει στην γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον από τον Φεβρουάριο εφέτος μετά από επιλογή του Γενικού Γραμματέα. Θα εγκαταλείψει λοιπόν τη γραμματεία μας και εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα ήθελα να του συγχαρώ και να του ευχηθώ του Μάικλ καλή τύχη σε αυτή την ε, τόσο σημαντική θέση για την σταθιοδρομία του και να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην γραμματή μας. Συγχαρητήρια Μάικλ Τόπιν. Τα πρακτικά Τις συνεδρίες της 10ης Δεκεμβρίου. Θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί εάν δεν υπάρξει μέχρι το τέλος της συνάντησης κανένα σχόλιο εκ μέρους σας. Σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες Πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού 1934 κάθετος 2006. Ο εισηγητής είναι ο συνάδελφος Χέλμουτ Σόλτς από την ΚΟΕ. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου Σόλτς Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην τελευταία συνεδρίαση των Προέδρων το θέμα αυτό ανεβλήθη και έτσι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Επίσης θα ήθελα να σας πω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας ότι στην τελευταία συνεδρία σας ενημέρωσα ότι είχαμε συνεννοηθεί για κοινό ε, χρονοδιάγραμμα με την ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Επίσης καθυστέρησε για να προετοιμάσει η ΑΦΕΤ το σχέδιο εκθεσής της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν την έκθεση 24 Φεβρουαρίου, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, εάν η ΑΦΕΤ αναβάλει, όπως φαίνεται για αργότερα, την ψηφοφορία και εμείς θα πρέπει να πράξουμε το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 15 Φεβρουαρίου, 5 το απόγευμα. Και κατά τη διάρκεια Τη συνάντηση των συντονιστών θα συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα της συμμετοχής μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή κυρίου Χέλμουτ Σόλτς για την παρουσία της έκθεσής του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαστε με αυτή την έκθεση ή που αναφερόμαστε στην έκθεση αυτή και ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και στους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους και επίσης τη γραμματεία και τον ε, κύριο Καλό ιδιαιτέρως οι οποίοι προσπάθησαν ε, να ε, διευκολύνουν την παρουσίαση του τεχνικού θέματος αυτού για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τεχνικά το μέσο αυτό. Ήδη τον Νοέμβριο είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και γι' αυτό δεν θέλω σήμερα να μακρηγορήσω. Ουσιαστικά έχουμε τρία ουσιαστικά θέματα κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να επεκτείνει γεωγραφικά την εφαρμογή του κανονισμού και ε, επ' αυτού θα πρέπει πλέον της ICI να ασχοληθούμε και με την DCI και αυτό είναι μία προσπάθεια την οποία προσπάθησα να τονίσω στην έκθεσή μου γιατί είπα ότι το ICI είναι το, το μέτρο, το κονδύλι το οποίο είναι ε, πιο αυστηρό και πρέπει να είναι ε, ελέγξιμο ιδίω σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας διότι με την συναπόφαση πολλά θέματα μπορεί να είναι αντικείμενο της εργασίας μας και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει ε, να ε, ε, δεν πρέπει, θα πρέπει να διευκολύνουμε την χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας σε πολλούς τομείς. Επίσης ε, όσον αφορά ε, την ε, οικονομική πτυχή αυτού του μέτρου θέλησα να, το, να την εξηγήσω και επίσης αναφέρθηκα στη νομική βάση ιδίως μετά τη μετάβαση στη συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες 24 και 25 που υπάρχουν στο κείμενο που έχω υποβάλει και όπου προσπαθώ με την βοήθεια της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατυπώσω μία μη ε, ε, ε, έκφραση για την εκτέλεση της εξουσιοδότησης διότι υπάρχουν ακόμη διαπραγματεύσεις για την τελική διατύπωση και πρέπει πρώτα να συνεννοηθούμε με άλλες επιτροπές και πλέον με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου δεν υπάρχει υπάρχει συνένεση για να εφαρμοστούν γενικώ ε, οι εκτελέσεις της εξουσιοδότησης παντού. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και αυτό ε, θα συζητηθεί και σήμερα το απόγευμα στη συνάντηση των συντονιστών. Θα ήθελα στο θέμα αυτό να αναφερθώ στο όνομα και στο μηχανισμό αυτού του εργαλείου και πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή θέλουμε ε, να ε, παραμείνουμε στη διατύπωση που υπάρχει όσα, όσον αφορά αυτό το μέτρο ή θα χρησιμοποιήσουμε ε, τη διατύπωση της Επιτροπής ΑΦΕΤ η οποία προσπαθεί να διατυπώσει πιο ευρέως αυτό το εργαλείο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα στην εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε εδώ και γι' αυτό θα ήθελα να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ε, τη διατύπωση ως έχει προς το παρόν. Ε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την κυρία Λόχ Μπίλε και να συνεννοηθούμε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Είπαμε ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί γρήγορα ή σχετικά γρήγορα αυτό το εργαλείο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα και μου ε, υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να διατηρήσει την 23η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία όπου θα ψηφιστεί η γνωμοδότηση στην ΑΦΕΤ οπότε να μπορέσουμε να σεβαστούμε το ισχύον χρονοδιάγραμμα. Οπότε ε, ούτως ή άλλως ε, το εργαλείο αυτό ε, θα εφαρμοστεί πια το καλοκαίρι και με τις καθυστερήσεις δεν ξέρω αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί καν το 2010. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει κατά την εξέταση ε, του σημείου αυτού. Ε, αυτά είχα να σας πω εγώ. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Το σχέδιο έχει ε, παρουσιαστεί και ξεκινώ με την ισκιώδη ε, ε, ε, συγγητρία την κυρία Γκότλιμπ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτς για την καλή συνεργασία καθότι επανειλημμένως συζητήσαμε την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι τελικά είναι πάρα πολύ καλό όλα τώρα να μπορέσουν να βασιστούν στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη νέα βάση ε, διότι δεν ήταν τόσο σαφή τα πράγματα στην αρχή τώρα όμως έχουν ξεκαθαριστεί και πιστεύω ότι μπορούμε γι' αυτό να συζητήσουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Αν καταφέρει η ΑΦΕΤ να σεβαστεί τις προθεσμίες της έχει καλός. Αλλά επειδή είμαι αναπληρωματικό μέλος και στην Επιτροπή αυτή. Δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί. Πιστεύω όμως ότι μετά από όλα όσα περάσαμε δεν χάλασε ο κόσμος αν έχουμε κάποια ακόμη καθυστέρηση για την εφαρμογή. Βέβαια καλό είναι να γίνει γρήγορα αλλά αν γίνει σωστά είναι πιο βασικό και έχω τρία σημεία να θίξω. Το πρώτο είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Στην αιτιολόγηση ε, όπου μιλάμε για τα επιπρόσθετα οικονομικά μέτρα ότι το μέτρο, το κονδύλι ICI θα χρησιμοποιηθεί στις υποανάπτυξη χώρες και δεν πρέπει να παρεμβληθεί στην ανάπτυξη. Αυτό είναι αμφισβητήσιμο διότι ξέρουμε ότι σε μία σειρά από υποανάπτυξη χώρες τα προγράμματα αυτά υιοθετούνται διότι ότι αυτά που θέλουμε να κάνουμε εκεί ε, δεν καλύπτουν άλλα κριτήρια. Αν λοιπόν γενικότερα ε, έχει να κάνει το θέμα με την ανάπτυξη νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και θα μπορούσαμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια και γι' αυτό πρέπει να εξαντλήσουμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό όσον αφορά την ε, τροπολογία 23 η οποία είναι πολύ πιο επουσιώδης από ότι το θέμα της χρηματοδότησης ε, ο εισηγητής θα ήθελε στην τροπολογία του να υπάρχει μία λεπτομερής ετήσια έκθεση και να υπάρχει υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέμα στο οποίο εγώ έχω μεγάλη πείρα για τις λεπτομερείς αιτήσει εκθέσεις. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε ούτε να τη διαβάσουμε σωστά είτε να την ελέγξουμε. Οπότε ή θα διαγράψουμε τον όρο λεπτομερής ή θα επεκτείνουμε την περίοδο, δηλαδή διετή περίοδο και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο γιατί έτσι όταν θα έχουμε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχουμε και το χρόνο και τη δυνατότητα να ψάξουμε τα πράγματα καλά και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο. Όσον αφορά το τρίτο θέμα, τον τριμερή διάλογο, η ΝΤΕΒΕ και η ΑΦΕΤ ήδη έχουν εμπλακεί σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και με εκπλήσει που από την αρχή δεν έχουμε συμμετάσχει ε, και εμείς σαν τρίτο μέλος και δεν πήγαμε δηλαδή και οι τρεις μαζί. Αλλά τώρα έχει αποκατασταθεί η κατάσταση και έτσι δεν θα ήθελα να πω εκ προημίου ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν θέλουν να συζητήσουν για τις εξουσιοδοτημένες ενέργειες διότι εις ε, την ε, συμφωνία σε ορισμένα θέματα οι απόψεις μεταξύ Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών ε, οργάνων διαφέρουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί εδώ πρόκειται για μία βάση εργασίας για τα επόμενα έτη και ε, ό,τι εμείς εγκαταλείψουμε τώρα δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν σωστά θυμάμαι, είναι η τρίτη φορά που συζητούμε την τροποποίηση αυτού του δημοσιονομικού μέσου του χρηματοδοτικού μέσου και νομίζω δεν πρέπει να προσθεθούν πολλά σε όσα ήδη υπόθηκαν. Εκτιμώ τη δουλειά του κυρίου Σόλτ και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους και οδησυσικητές και τις ομάδες τους για να καταλήξουμε σε ένα συνεργατικό κειμένο και να καλύπτουμε όσο δυνατόν περισσότερο του στόχου μα. Νομίζω ότι ω τώρα μπορούμε να έχουμε θετική αποτίμηση του έργου μα και μάλιστα στο χρονικό διάστημα που μα διατέθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η έκθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μα με την Επιτροπή ΑΦΕΤ, καταλαβαίνω και τι δικέ του απαιτήσει, αλλά αυτό αφορά περισσότερο τι διαθεσμικέ, τι εσωτερικέ σχέσει του Κοινοβουλίου, δηλαδή των Επιτροπών μεταξύ του. Εμείς δεν μπορούμε να αποφανθούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά την ουσία. Θα συμφωνήσω με την εκκλήση κυρίου Σόλτς για το θέμα της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι είναι θεμελιώδους σημασία. Πολύ σωστά η Επιτροπή σκέφτηκε να, να διευρύνει τον κανονισμό ώστε να καλύπτονται και άλλες χώρες. Ο κόσμος μας αλλάζει και μάλιστα ραγδαία και Υπάρχουν στον κόσμο χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται στην, στον δρόμο της ανάπτυξης βεβαίως, αλλά και άλλες αναδυόμενες οικονομίες και μάλιστα με αρκετή ορμή στην παγκόσμια αγορά. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και αυτό ενδιαφέρει και τα στρατηγικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε άλλες χώρες, στο εσωτερικό των ίδιων χωρών που προηγουμένως ανέφερα, υπάρχουν και καταστάσεις φτώχειας τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να ενισχύσουμε, να τις καταπολεμήσουμε δίνοντας κονδύλια. Είμαστε ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της ε, αναπτυξιακής βοήθειας στον πλανήτη, αλλά αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα και να καμαρώνουμε γι' αυτό, δεν μπορούμε παρόλα αυτά να παραμερίσουμε και τις βιομηχανικές, οικονομικές και πολιτικές ε, σχέσεις και διασυνδέσεις που είναι ο στόχος αυτού του κανονισμού. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε επιπλέον πολιτικές και να στοχεύσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις πέραν αυτού του κανονισμού. Αυτή είναι η πρώτη μου βασική παρατήρηση. Το θέμα είναι λοιπόν και γενικότερα πολιτικό, όχι απλώς οικονομικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση περί τούτου. Πάντως, Σωστά εδώ σταθήκατε και στο ρόλο του Κοινοβουλίου σε σχέση με το όλο θέμα. Και σε σχέση με την παρέμβαση της κυρίας Γκότλιμπ και σεβόμενος βεβαίως τις ιδέες της, παρόλα αυτά να θυμίσω ότι εμείς είμαστε εκείνοι που οφείλουμε να φροντίζουμε η συνθήκη της Λισαβόνας να ισχύει για το δημοκρατικό και νομοθετικό βίο της Ευρώπης κατά τον τρόπο και το πνεύμα όπου συνελήφθη η συνθήκη αυτή και κατά τον οποίο εγκρίθηκε. Αυτά όλα απαιτούν εντατικέ προσπάθειες από την πλευρά και των άλλων θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ένα στοιχείο είναι οι διαθεσμικές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων, αλλά κάποιες φορές δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά ως ε, έναν επιπλέον κόπο, μια ταλαιπωρία στις στενές σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Και εδώ να πω στον κύριο Σόλτ, ότι δεν ξέρω αν ο σωστό όρο είναι εδώ λεπτομερή εντελεχή ή κάτι άλλο, αλλά το να αναζητούμε, πρέπει να το επισημάνω αυτό, το να αναζητούμε μια ενισχυμένη σχέση, μια στενότερη σχέση με το εκτελεστικό, κατεξοχήν εκτελεστικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει και το δικαίωμα τη νομοθετική πρωτοβουλία, μου φαίνεται ότι αυτό πραγματικά είναι καθοριστική σημασία για τι διαθεσμικέ μα σχέσει. Και είναι και κάτι που ε, βασίζεται και απορρέει και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλουμε λοιπόν σχέσεις πολύ πιο στενές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις γενικόλογες απαντήσεις που συνήθως λαμβάνουμε όταν τις υποβάλλουμε ερωτήσεις. Και το τρίτο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι οι τροπολογίες 10 και 11 που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ρόλο που μπορούν να αναλάβουν στη διεθνή οικονομική συνεργασία είναι σωστές. τι ημεριζόμαστε. Απλώς για την τροπολογία 5 στο τέλος των παρατηρήσεών μου ήθελα να πω ότι έχω την εξής εντύπωση. Σήμερα νομίζω ότι μοιάζει να διευκρινίζει η τροπολογία αυτή. Το κείμενο τελικά οδηγεί σε σύγχυση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενεργήσει, να αναλάβει δράση και αυτό στο πνεύμα των θεμελιωδών αρχών της. Αυτό ίσω να φαίνεται προφανέ, αλλά είναι μια έκκληση που πάντοτε πρέπει να γίνεται. Ταυτόχρονα είναι προφανέ ότι ο κατάλογος ο πρόσθετο κατάλογο των επιπλέον χωρών που θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, ο κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνει χώρε με τις οποίες εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα μπορούσα να πω ότι συμμεριζόμαστε και έχουμε τι ίδιε αξίε, τι ίδιε θεμελιώδει αξίε. Μπορεί όμω να έχουμε κοινά στατηγικά συμφέροντα. Το να μην έχουμε τίποτα κοινό με συστήματα και αρχέ που διέπουν την λειτουργία του κράτου τη Κίνα σήμερα είναι ένα στοιχείο. Ίσως να υπάρχει ένα γενικό αίσθημα ανθρώπινης επαφής με τα πρόσωπα όμως και με τους πολίτες, όχι με το καθεστώς. Και αν σκεφτούμε και τις άλλες 150 χώρες στον κόσμο, ε, που είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν φιλελεύθερη οικονομία, ούτε δημοκρατικά πολιτεύματα απαραίτητο. Συστήματα που δεν συνάδουν με την ε, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αυτά, δεν μπορούμε, με τα κράτη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα κοινά. Και να πω και κάτι ακόμα. Εμεί όταν βρούμε, όταν ενεργούμε και όταν χρηματοδοτούμε, θέλουμε ω αντάλλαγμα να υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τουλάχιστον βελτίωση του, της προστασίας τους των αρχών που διέπουν ε, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η χάρτα των θεμελιωδών ε, ε δικαιωμάτων στο άρθρο της 212 θυμίζει και τον κανονισμό του 2004 που τον τροποποιεί και όλα αυτά μας δίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για να πούμε ότι το παρόν κείμενο της Επιτροπής θα μπορούσε και όσοι έχει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω τροπολογίες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ απλώ να σα επισημάνω ότι έχουμε ένα μακρύ κατάλογο θεματών που θα πρέπει να συζητηθούν. Γι' αυτό θα σα παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Κύριε Αρνέζ δεν είναι εδώ. Εκπρόσωπος των Πρασίνων δεν είναι εδώ. Κύριε κύριος από την ε, ΦΔΑΡ, όχι. Τότε ο πρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Έχω μια γενική ανησυχία για ε, την, πολιτική διάσταση που λαμβάνει η εμπορική μας πολιτική. Είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και θεωρούμε ότι αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και ότι επιτρέπει και στον κόσμο μας να γίνει ένα καλύτερο μέρος. Το χρηματοδοτικό λοιπόν μέσον για να ενισχύσουμε τι εμπορικέ σχέσει προφανώ είναι κάτι που μα βρίσκει σύμφωνο. Απλώ αυτό που μα ανησυχεί είναι η εμπορική διάσταση που λαμβάνει η εμπορική πολιτική. Γνωρίζω την ε, ε, ανησυχία της ε, Βαρόνης Άστον, της συναδέλφου μου, και πρέπει να σταθώ εδώ στην τροπολογία 2 για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα βασικά δικαιώματα και την τροπολογία 5 όπου η Ένωση θέλει να προωθήσει τις αρχές της. Αυτά όλα ανησυχούν τη συνάδελφο και να πω ωστόσο ότι όλοι έχουμε αξίες, όλοι είμαστε δημοκράτες, όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο. Όμως γνωρίζουμε ότι σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να τα εξετάσει κανείς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Και εδώ να θυμίσω και τον πρόεδρο Τσάβες της ε, Βενεζουέλα. ο οποίο θεωρεί ότι είναι μεγάλο υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρόλο που καταπιέζει τι βασικέ ελευθερίε των πολιτών του. Η δική μου λοιπόν άποψη είναι ότι το να δίνουμε πολιτική διάσταση σε ένα μέσο όπως αυτό που είναι χρηματοδοτικό ε, είναι ενσφαλμένο, διότι θα πρέπει να έχει τεχνικό χαρακτήρα εξέταση του θέματος. Δεν αναζητούμε εδώ τρόπο να προωθήσουμε τις πολιτικές ατζέντες συγκεκριμένων προσώπων και πολιτικών. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά αυτά που ακούω είναι απαράδεκτα. Εάν το να ασκεί κανείς την πολιτική Σημαίνει ότι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμό των δικαιωμάτων των συνδικαλιστών, ο ε, σεβασμό των... Ε, και προστασία των παιδιών και ούτω καθεξής εάν αυτό είναι λάθο, τότε πάμε να είμαστε πολιτικοί. Όχι, γιατί εάν η φτυχία του Άγγλου καταναλωτή πρέπει να πληρώνεται με τη δυστυχία ανθρώπων, ε, γυναικών και ανδρών σε όλο τον πλανήτη, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε επάγγελμα ίσω. Σίγουρα σε αυτή την περίπτωση να ξέρει ο συνάδελφο ότι δεν συμμεριζόμαστε τι ίδιε αξίε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριο Γκάρι Μίλλερ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Γκάρι Μίλλερ από την Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε εδώ το σχέδιο έκθεση του κυρίου Σόλτ και τον ευχαριστούμε για το επικοδομητικό πνεύμα με το οποίο Εξέταζε το θέμα και τη στενή συνεργασία που είχε μαζί μας. Το εκτιμούμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Απλώς να περιοριστώ στο εξή. Σε δύο σημεία. Πρώτον, στην Επιτροπή ανησυχούμε κάπως για το χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε, ο στόχο του μέσου αυτού είναι να χρηματοδοτήσει κάποια προγράμματα που ξεκινούν από το εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στι χώρε που αναφέρονται στο κατάλογο. Και όπου θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι δεν μπορούμε πια να τα χρηματοδοτήσουμε με το μέσο ανάπτυξη. Αυτά τα προγράμματα θα αρχίσουν να χρηματοδοτούνται από του χρόνου, από τον Ιανουάριο. Αλλά το χρονοδιάγραμμα αυτό κάπως μας ανησυχεί, γιατί τα βασικά έγγραφα για τον επόμενο χρόνο πρέπει να ετοιμαστούν εγκαίρως. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της έκθεσης είναι κάτι που θα το προλάβετε, θα το τηρήσετε. Και η Επιτροπή θα εξυπηρετήσει όσο μπορεί τον κύριο Σόλτ και την Επιτροπή σας να πετύχει τους στόχους της. Απλώς για τις τροπολογίες του κύριου Σόλτ είναι αρκετές τι έχουμε εξετάσει προσεκτικά στην Επιτροπή. Τα συζητήσαμε με τον κύριο Σόλτ επίση. Και δεν θέλω εδώ να περάσω σε λεπτομέρειε για τι τροπολογίε ξεχωριστά. Αλλά είμαστε στη διάθεση του κυρίου Σόλτ και τη κυρία Λακμπέρεντ στην ε, ΑΦΕΤ ώστε να πετύχουμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο εν ώψη των ψηφοριών σα, ώστε να επιταχυνθεί και όλη η διαδικασία. Να έρθω στο δεύτερο βασικό ζήτημα που ήθελα να θίξω, η επιτροπολογία. Οι εκπροσώποι τη Επιτροπή νομίζω το έχουν αναφέρει ξανά αυτό στην Επιτροπή σα, να επαναλάβω στη θέση μα. Είναι σαφέ ότι εδώ έχουμε διαφορετικά νομικών, διαφορά νομικών απόψεων μεταξύ Επιτροπή και Συμβουλίου, αλλά και Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ακολουθεί την ίδια προσέγγιση σε όλε τι επιτροπέ και σε όλε τι εξωτερικέ σχέσει. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το δούμε κατά τρόπο οριζόντιο. Αναφέρεται ότι επίκενται συζητήσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων σύντομα, ένα τριμερή διάλογο, αλλά δεν θέλω εδώ να αναλύσω τι διαφορέ απόψεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Πρόεδρε. Γνωρίζω, φαντάζομαι μάλλον ότι περισσότεροι τα γνωρίζουν αυτά. Η Επιτροπή θεωρείται τα στατικά έγγραφα που εγκρίνονται από την ίδια για το μέσο αυτό, όπω και άλλα, δεν μπορούν να θεωρούνται delegated acts, δηλαδή εξουσιοδοτημένε πράξει κατά εξουσιοδότηση. Δεσμεύουν συγκεκριμένα πρόσωπα και εδώ φαίνεται να υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του συγκεκριμένου άρθρου της συνθήκης που προβλέπει τη νέα αυτή έννοια των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί η κατάλληλη διατύπωση και για τις τροπολογίες που περιλαμβάνει η έκθεση. Από την άποψη της Επιτροπής πάντως να πω Αυτό που είπε αυτό που είπε η συναδελφό σα ότι αποφεύγουμε το θέμα αυτό διαρκώ είναι κάτι που δεν ισχύει. Θέλουμε να συζητηθεί το ζήτημα, θέλουμε να βρεθεί λύση. Και ελπίζουμε να συμβεί αυτό. Και γι' αυτό θα συμμετάσχουμε και στον τριμερή διάλογο με τρόπο ενεργό. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την επίτευξη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Επιτροπή βεβαίω για το θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε, και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την ε, στενή συνεργασία με τον κύριο Σόλτ, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν τι προφορίε του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φαίνεται να μην υπάρχουν μόνο διαφορέ απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά και μεταξύ των μελών τη ίδια μα τη Επιτροπή. Ο κύριο Σόλτ τώρα για να κλείσει η συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, για τις υποδείξεις ε, και για τα σχόλια από τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία σημεία. Προσπάθησα να ε, να ε, διευκρινίσω ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους επιζητούμε και βεβαίως έχουμε στρατηγικά συμφέροντα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ε, θέματα που είναι ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικονομικά δικαιώματα να μπορέσουν να προωθηθούν στις χώρες με τις οποίες έχουμε συναλλαγές. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα αυτή τη διατύπωση. Πρέπει να ξαναδώ το αγγλικό κείμενο. Το γερμανικό είναι αρκετά σαφές. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι προσπαθούμε ε, εδώ να αναφερθούμε σε στρατηγικά συμφέροντα αλλά να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους θέλουμε να συνεργαστούμε. Ε, στη συνέχεια θα πρέπει ούτως ή άλλως να συμφωνήσουμε στο επίπεδο των συντονιστών όπως είπα διότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ της ε, Επιτροπής του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και ακόμη εντός του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ε, εγώ θα ήθελα να πω τη γνώμη μου σαφώς. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία εμπλοκή ε, του Κοινοβουλίου εις τις εντεταλμένες νομικές πράξεις και ε, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και να προσπαθήσουμε μέσω διαπραγμάτευση να καταλήξουμε σε μία αποδεκτή λύση ε, ε, και εμένα με ενδιαφέρει το θέμα αυτό οπότε αν όλοι οι συμμετέχοντες και στις επιτροπές ενδιαφερθούν θα προσπαθήσω με την με τις άλλες επιτροπές ε, να συνεργαστώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ε, του εργαλείου αυτού και να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Με αυτά κλείνει η συζήτηση. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 15 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 16 και 17 Μαρτίου. Τώρα ας προχωρήσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, εξέταση του σχεδίου έκθεσης, που είναι δική μου. Όπως τα γνωρίζετε, η πρόταση της Επιτροπής αρχικά απεστάλλει στο Κοινοβούλιο βάσει της διαδικασίας διαβουλεύσεων αλλά δεδομένων των αλλαγών που προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή μας, επισχέθη, μας στην προηγούμενη συνάντησή μας ότι η επικοινωνία μεταξύ μας θα αλλάξει κατά τρόπο ώστε η νομική βάση για την έγκριση της πρότασης αυτής να βασιστεί στο άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα έχουμε την επίσημη νομοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου αυτού. Όμως, εξ όσων γνωρίζω, η αλλαγή αυτή ακόμη δεν έχει επέλθει. Έχουμε όμως την υπόσχεση της Επιτροπής. Αυτές οι επίσημες διαδικασίες και τυπικότητε μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο. Έτσι λοιπόν, ετοίμασα το σχέδιο έκθεσης προκειμένου να λάβω υπόψη τα σχόλια της ε, πρώτης συζήτησής μας. Εδώ στηρίζω την πρόταση για τις διατάξεις χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, διότι είναι μια σημαντική χώρα και σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται τη συνδρομή μας. Ωστόσο, στην πράξη, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πρόσθετη δανειοδότηση 500 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί από την Επιτροπή. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις από την Ουκρανική πλευρά. Όπω θα διαβάσετε και στην έκθεση της Επιτροπής, στην πρόταση μάλλον τη Επιτροπή, ω τώρα, ακόμη και τα 110 εκατομμύρια ευρώ συνδρομής που δόθηκαν το 2002, δηλαδή πριν 7 χρόνια, δεν έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Διότι η Ουκρανία δεν έχει καλύψει τις βασικές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί τότε. Έτσι λοιπόν προτείνουμε τα κονδύλια αυτά να διατεθούν αργότερα. Για να εκταμιεύσει το δάνειο αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει αυστηρότερε ε, προϋποθέσεις. Συνολικά για την οικονομική συνδρομή το πρόβλημα είναι ότι εμεί στο Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουμε ποιε θα είναι παλιέ προποθέσει προϋποθέσεις ή άλλως και ποιε θα είναι οι νέε που προτείνονται. Θα δείξουμε εμπιστοσύνη βεβαίω στην γνώση τη Κομισιόν για τα θέματα αυτά, όμω επίση γνωρίζοντα ότι η Επιτροπή χρειάζεται περιθώριο ευελιξία ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί τι σχετικέ συμφωνίε και να δώσει συνδρομή. Πρέπει να του το επιτρέψουμε αυτό. Και εμεί βεβαίω δεν μπορούμε να αναλάβουμε το ρόλο τη Επιτροπή εδώ και να θέσουμε τι βασικέ προποθέσει στη θέση τη. Όμω θα πρέπει να υπάρχει υπόλογο για την προτινόμενη οικονομική συνδρομή και να είμαστε βέβαιοι ότι θα βελτιωθούν οι προποθέσει, η αυστηρότητά του τουλάχιστον, χωρί να πληγεί η αγορά και η εμπορική μα πολιτική. Επίση, έχω υποβάλει αρκετέ τροπολογίε προκειμένου να ισχυθεί ο ρόλο του Κοινοβουλίου σχετικά και να βελτιωθεί και ο τρόπο που έχουμε ενημέρωση για τα ζητήματα αυτά. Έχετε το σχέδιο έκθεση μπροστά σα, δεν χρειάζεται να προχωρήσω σε λεπτομέρειε. και να εξηγήσω τις, λεπτομέ... τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες, να δώσω το λόγο στους χειώδεις εξηγητές. Από την ομάδα του ΕΛΚ, ο κύριος Κουίγκλερ. Ε, uh, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο στο θέμα αυτό. Δηλαδή θα χρειαστούμε δύο-τρεις μήνες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω την καλή συνεργασία που είχα με τη Γραμματεία ε, για την κατάρτιση της γνωμοδοτήσεώς μας. Είδα τις τροπολογίες σας κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλές και θα ήθελα να τονίσω ορισμένα θέματα. Δηλαδή Καταρχήν, στην επεξηγηματική δήλωση ότι αναφερόμαστε στην Ουκρανία όχι μόνο σαν στρατηγικό συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και δυνητικό μελλοντικό ε, υποψήφιο μέλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια το θέμα είναι πολιτικό και εδώ δεν θέλω να ξεκινήσω ε, μία συζήτηση αλλά πιστεύω ότι οι αξίες μας θα πρέπει να είναι προσιλωμένες σε ε, οικονομικά και κοινωνικά θέματα αλλά συγχρόνως να προασπίζουν την σωστή χρηστή διακυβέρνηση κυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε έρχομαι εις ε, την τροπολογία για τους όρες οι οποίοι, ε, από τους οποίους θα εξαρτάται η χρηματική βοήθεια και συμφωνώ ότι πρέπει να αυξηθεί και η διαφάνεια και ε, η ε, ευθύνη και πιστεύω ότι δεδομένες καταστάσεις ε, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή δηλαδή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα στην περίπτωση της Ρουμανίας πρέπει να σας πω ότι οι έντονες συζητήσεις οι οποίες συνδυάζονται με οποιαδήποτε συμφωνία ισχύουν και για τα κράτη-μέλη και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οπότε το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της ε, αποδόσεως λογαριασμών, το θέμα της ε, βοηθείας και της ε, χρήσης της βοήθειας είναι διάφορα θέματα ε, συνδεδεμένα μεταξύ τους και ε, που ε, αναφέρονται σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου συζητούνται αυτή τη στιγμή έντονα και η διαφάνεια, η απόδοση λογαριασμών, όλες οι συζητήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για να θέσουμε τους όρους και την εξέλιξη των όρων για να δούμε εάν όντως οι όροι αυτοί, οι προϋποθέσεις αυτές επί της ε, συγκεκριμένης περιπτώσεως στην ε, Ουκρανία επιτρέπουν να χορηγήσουμε αυτή τη βοήθεια. Είναι κάτι που χρειάζεται, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο για να αυξήσουμε τη διαφάνεια στις χώρες αυτές. Και τέλος, σχετικά με την ίδια ιδέα, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση και ε, την χρησιμοποίηση αυτών των πόρων, είναι θέματα με τα οποία συμφωνώ πλήρως. Είναι παρόντες οι υπόλοιποι σκιώδεις συζητητέ. Αν κανένα άλλο λοιπόν δεν θέλει να συμμετέχει στη συζήτηση, κοιτάξτε. Μία ερώτηση για κάποια λεπτομέρεια που αφορά την Κομισιόν. Ίσως να μου απαντήσει γραπτό γιατί δεν έχουν χρόνο. Λέγεται ότι η Επιτροπή στην αιτιολογική ε, έκθεση ότι θα χορηγήσει αυτή την μακροοικονομική βοήθεια μέχρι 500 εκατομμύρια ευρώ πράγμα που θα επιτρέψει το ποσό αυτό ή να το δανειστεί από τις κεφαλαίες αγορές ή από τις διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. οι χώρες που είναι οι, χώρες που συνεισφέρουν θετικά στον κοινωτικό προϋπολογισμό θα κληθούν να καταβάλουν κάποιο ποσό. Ποιος είναι ο μηχανισμός που θα ακολουθήσει η Επιτροπή για τη χορήγηση αυτών των 500 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη συνήθεια διαδικασία αλλά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Δερμιτζιώτη για να δώσει μια απάντηση στο σχόλιο αυτό και να ε, σχολιάσει και την εταιρεία έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ πολύ διότι προετοιμάσατε πάρα πολύ έγκαιρα την έκθεσή σας με την κατάθεση τροπολογιών. Είναι πολύ χρήσιμα, επικοδομητικά. Υπάρχουν τριών ειδών τροπολογίες. Τροπολογίες που αφορούν την νομική πτυχή του όλου θέματος, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχει καλός. γίνεται αναφορά στη νέα συνθήκη, στα νομικά θέματα και γίνεται και αναφορά στις θεσμικές αλλαγές που έχουν σχέση με τη νέα συνθήκη. Οι δύο τελευταίου τύπου τροπολογίες είναι τροπολογίες τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Σας ευχαριστούμε. Αλλά επαναλαμβάνω για τους δύο τελευταία είδη τροπολογιών αυτήν ε, τη στιγμή ε, δεν έχουμε ακόμη τη νέα επιτροπή τα θέματα λοιπόν πολιτικής ακόμη δεν μπορεί να τα χειριστεί θα θέλαμε όμως να συνεργαστούμε με εσάς επικοδομητικά και με το Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μία λύση συμβιβαστική θετική που θα μπορέσει να σα οδηγήσει σε ένα κείμενο αποδεκτό από όλου. Διότι πρόκειται σύμφωνα με τη νέα συνθήκη για την πρώτη περίπτωση που αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο πιο θετικός και επιδεικνωμένος τρόπος να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από όσον κατάλαβα δεν μου ζητάτε να σχολιάσω λεπτομερώ τι διάφορε τροπολογίες. Για να απαντήσω τώρα την ερώτηση για το uh, για το Omnibus Act της Κομισιό στις ε, επόμενες μέρες θα υπάρχει τροπολογία της προηγούμενης πράξης και ελπίζουμε ότι θα την ε, έχει διαθεσή σας σύντομα εκτιμούμε το γεγονός ότι αρχίζετε να εργάζεστε για το όλο θέμα πριν να έχετε ακόμη και την επίσημη πρόταση της ε, Κομισιόν και θα μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε, ελπίζω, σε ένα κείμενο που θα ικανοποιεί τους πάντες. Τώρα, στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε, όντως, δεν πρόκειται για δάνειο που προέρχεται από τον ποσό, που προέρχεται από τον κοινοτικό προπολογισμό, προσφεύγει στις αγορές, δανείζεται η Κομισιόν και δανείζει την χώρα, χορηγεί το κονδύλι αυτό στη χώρα. Δεν πρόκειται λοιπόν, αν θέλετε, για κοινοτικά χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε μια ειδική χώρα. Υπάρχει λοιπόν εμέσως ε, ε συνεισφορά της Κομισιόν στα πλαίσια του μηχανισμού εγγύσεων. Άρα δεν υπάρχει καμία άμεση, αν θέλετε, επίπτωση για τον κοινοτικό προβλήμα. Δεν είναι κοινοτικά τα κονδύλια. Το ερώτημα αφορούσε τους μηχανισμούς και ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο, αν προβλέπεται κάποιο επιτόκιο. Κατάλαβα ότι δεν προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια. Έτσι όμως χορηγεί η Κομισιόν χρήματα δεν προέρχονται από τα δικά τη ε, κονδύλια. Και επειδή με ενδιαφέρει τι πληρώνουν οι Άγγλοι φορολογούμενοι, θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι λεπτομερό ο μηχανισμό. Αν θέλετε να μου δώσετε λεπτομερή απάντηση γραπτός. γραπτός. Για μας και βεβαίως και για τους υπολείπους συναδέλφους. Νομίζω ότι και πολλά άλλα μέλη της Επιτροπής μας θα ενδιαφέρονταν για την χορήγηση χρημάτων σε κάποιους και κονδυλίων αν δεν τους κοστίζει τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν μπορεί να βρει τέτοιο μηχανισμό η Κομισιό ε, που δεν μας κοστίζει τίποτα σε όλους εμάς θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε γραπτός για με λεπτομέρειες πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας στείλουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον όλο Τώρα, εάν ε, θέλετε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Επιτροπή προσφεύγει στις κεφαλαιαγορές, δανείζεται, συνήθως με, σαν ε, δανείζεται ομολογίες, ομόλογα. Όσον αφορά το επιτόκιο, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με ενδείξεις που είχαμε τις διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται τα θέμα αυτό, πρέπει να σας πω ότι το επιτόκιο που αφορά αυτά τα ποσά είναι της τάξης του 4%. Το κόστος ε, βεβαίως δεν βαρύνει εμάς, βαρύνει την Ουκρανία τα ε, χρήματα αυτά θα καταβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ουκρανία και θα τα καταβάλει στους επενδυτές ε, μετά η Κομισιό. Οι επιπτώσεις ε, για τον προϋπολογισμό περιγράφονται σε διάφορα σχετικά έγγραφα τα οποία εσύ συνάπτονται, αλλά ούτως ή πάλως υπάρχει η υπαρχει η εγγυηση για αυτά τα κονδύλια τα οποία καταβάλλονται σε τρίτες χώρες από την Κομισιόν. Η δάνεια Euratom, η μακροοικονομική βοήθεια, και βεβαίως εδώ το επιτόκιο είναι της τάξης του 9% αλλά με διαφορά. Με κάποια καθυστέρηση. Γίνονται προβλέψεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και εάν υπάρχει κάποια διαφορά καλύπτεται από μια γραμμή του προϋπολογισμού. Συνήθως ε, υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για να μπορέσουν να καταβληθούν αυτά τα ποσά αν υπάρχει διαφορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας στείλουμε πιο ε, γραπτός περισσότερα σε εξηγήσει σε σχέση με τον όλο μηχανισμό. Σας ευχαριστώ. Μας επεξηγήσετε κάποια τα πράγματα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε γραπτός τις πληροφορίες για το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλια τα οποία κάνατε, για το σχέδιο εκθεσής μου. Πρέπει να σας πω ότι έκανα την έκθεσή μου πάρα πολύ γρήγορα, χάρη στην πολύτη βοήθεια της γραμματείας του Μάρκ, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μπόρεσα λοιπόν να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης και θα κάνω την ε, τελική μου έκθεση. Σύντομα λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια που έκανε και ο συνάδελφος του ΕΛΚ και όπως είπε και η Επιτροπή θα προσπαθήσει στο τέλος να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι ικανοποιητικό για τους πάντες. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 15 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 16-17 Μαρτίου εφέτος. Ευχαριστώ. Περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία. Σχέδιο γνωμοδότησης. Δίνω το λόγο στην συντάκρια Μαρία Μουνής Δεουρκίθα. Απλώς θα ήθελα να πω ότι Πεφάσισε η Επιτροπή ΔΕΒΕ να συντάξει την έκθεση και εμείς απλώς συντάσσουμε γνωμοδότηση επί αυτού του θέματος. Βλέπουμε να υπάρχουν ε, κάποια σημάδια οικονομικής ανάπτυξης για κάποιες χώρες. Υποφέρουν όμως εξαιτίας οικονομικής κρίσης ακόμη οι αναπτυσσόμενες χώρες και εξαιτία της οικονομικής ύφεσης υπάρχουν ακόμη προβλήματα και με τις ε, ε, άμεσε επενδύσει και με άλλα θέματα. Η Μαρία Μουνίχη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Όπω είπα και στι προηγούμενε παρεμβάσει μου, μία από τι επιπτώσει οικονομικής κρίσης είναι ότι έχουν μειωθεί τα οι έσοδα από εξαγωγές στις αναπτυσσόμενες χώρες, πράγμα το οποίο απειλεί να καταστρέψει την ε, οικονομική ε, βελτίωση και την ανάπτυξη των νότων. Ο κύριος Ενρίκε Γκερέρο έχει συντάξει τη σχετική έκθεση και εγώ στη δική μου γνωμοδότηση θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στις αναπτύξεις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη των αναπτυσσομένων ε, χωρών ουσιαστική. Και θα ήθελα να ληφθούν υπόψη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας και η μείωση των τιμών καταναλωτή. Θα ήθελα τελικά να υπάρξει ε, πολύ καλή ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα το 2010 για να μπορέσει να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη από την κρίση έτσι όπως είχε γίνει και με τις χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να μειωθούν οι τιμές καταναλωτή. Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η στρατηγική της βοήθειας στο εμπόριο έχει ως στόχο να στηρίξει αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να αρχίσουν να επωφελούνται από τις οικονομικές συμφωνίες, να διευρύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και να επιταχύνουν την εξάλληψη το Ζητείτε από την Επιτροπή λοιπόν να εξασφαλίσουν την καταβολή των πιστώσεων και τους ζητούμε να υποστηρίξουν τις ε, ε του εμπορίου στις, με χώρες μεταξύ νότου-νότου. Η τροπολογίες έχουν ε, ήδη κατατεθεί. Οποιαδήποτε σχόλιο εκ μέρους των συναδέλφων είναι καλόδεχθες για να μπορέσει να βελτιωθεί η έκθεση τελικά. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Ζήτησαν το λόγο κάποια μέλη της Επιτροπής και μετά θα δώσω τον λόγο στην Επιτροπή. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, εν ονόματι του Κρίσιαν Όμπο, ο οποίο έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ευχαριστώ για το σχέδιο που μας έχει υποβληθεί. Συμφωνούμε με τα περισσότερα θέματα. Ευχαριστούμε για την ισοσκελισμένη παρουσίαση. Θα κάνουμε ορισμένε τροπολογίες για να βελτιώσουμε τη διατύπωση, αλλά προς το παρόν σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και για το σχέδιο που παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Ντάνιελ Κασπάρη σχετικά με το τι έχει γίνει. Νομίζω ότι έχετε καλύψει τα περισσότερα θέματα που επιθυμούσαμε και νομίζω ότι είναι μια ισοσκελισμένη έκθεση. Βεβαίως υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα όπου πρέπει κανείς να αναγνωρίσει το ρόλο των τραπεζών αλλά και την έλλειψη εποπτείας. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι οδήγησε στην οικονομική κρίση γιατί υπάρχουν και θέματα πράγματα που δεν ε, κατάλαβαν οι ρυθμιστές ε, που δημιούργησαν την κρίση και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σε πολλές από τις χώρες αυτές ε, δεν υπάρχει καμία πρόοδος διότι ακόμη οι χώρες που έχουν απελευθερωθεί μετά από 40 χρόνια υποφέρουν από τις παλιές πολιτικές και είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε. Δεν είναι κάτι απλό ε, δεν φτάνει να ε, επικρίνουμε τις τράπεζες, πρέπει να εξετάσουμε και τη νομική πτυχή. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να αναφερθώ εις ορισμένα θέματα της, ε, του σχεδίου της γνωμοδότησης ε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό να υπάρχει μία πιο συνεκτική πολιτική και να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάπτυξη από τη μία μεριά αλλά υπάρχει και το εμπόριο από την άλλη και πρέπει να δούμε ότι το εμπόριο ε, μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της φτώχειας ε, πρέπει να στηρίξουμε και τους ε, ε, επιχειρηματίες. Όταν προσπαθούμε λοιπόν να μιλήσουμε στους επιχειρηματίες, όταν επισκεπτόμαστε αυτές τις χώρες, μας μιλούν για τις πολιτικές της Ευρώπης και παραπονούνται, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις δικές τους πολιτικές και ε, αν έχουν χρήματα κοιτάζουν ε, να τα επενδύσουν και να έχουν καλύτερες θέσεις αλλά ε, δεν θα αγοράσουν γη παραδείγματο χάρη γιατί δεν ξέρουν αν την επόμενη το πρωί θα την έχουν ακόμη Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ οι τοπικοί επιχειρηματίες, ο ρόλος τους, η κοινωνία των πολιτών ε, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν αλλά έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή αυτή την τελευταία τετραετία. Νομίζω ότι ε, και η δεξιά πτέρυγα και η αριστερή του Κοινοβουλίου θέλουν να λύσουμε το πρόβλημα του προστατευσιμισμού και θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τις φτωχές χώρες ε, από τον ανταγωνισμό των πιο πλουσίων χωρών. Η Γκάνα παραδείγματος όταν ε, ε, ε, εξάγει το ε, ε, το ε, μεγαλύτερο ποσοστό των, της παραγωγής της σημαίνει ότι στην εισαγωγή είναι υψηλή οι δασμοί και ακόμη και οι φτωχοί δεν μπορούν να πληρώσουν τους δασμούς για είδη που τους είναι πρώτης ανάγκης. Άρα οι δασμοί είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να ισχύσει μακροπρόθεσμα. Μιλήσατε για την κεφαλοποίηση ορισμένων τραπεζών. Πέρυσι μιλούσαμε επιχειρηματίες από την Αυτική και τους ρωτούσα τι θέλετε από μας, τι θέλετε το οποίο μπορούμε να σας ε, προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά τι άλλα θέματα υπάρχουν και μας είπαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει το σωστό πλαίσιο, οι σωστοί κανονισμοί, οι σωστοί νόμοι για τις παροχές όχι μόνο δηλαδή τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, αλλά και ιστοσελίδες και άλλα θέματα που επηρεάζουν πάρα πολύ διότι υπάρχει ε, μία ιστοσελίδα η οποία επιτρέπει να γράψει κανείς στους επιχειρηματίες στις χώρες αυτές και ζητούν επίσης να γίνουν περισσότερες τράπεζες και ένας παραγωγός, ένας κοινοτρόφος που ε, είχε χρειαζόταν χρηματοδότηση ε, και μας ζητούσε ιδεολογικά κάνα να υπάρχει μεγαλύτερη πολυμορφία χρηματοδότησης. Ε, υπάρχουν λοιπόν διάφορα είδη παρόχων χρηματικής ενισχύσεως που θα έπρεπε να αναπτυχθούν. Ο εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε επειδή επικαλύπτεται το θέμα αυτό με το επόμενο που αναφέρεται ή στην ε, συνοχή της πολιτικής πιστεύω ότι εδώ ζητείται μια συνεκτική πολιτική και μια συνεργασία με τις ανάπτυξη χώρες αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ αυτού που λέγεται εδώ και ε, της ε, του γύρου της Ντόχα και της οικονομικής ε, διαδικασίας η οποία πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα της ε, ε, φτώχειας κατ' εμέ η διαδικασία του ΠΟΕ έχει επηρεαστεί από την κυριαρχία των πιο ε, ισχυρών οικονομικών μπλοκ διεθνώς που δεν ενδιαφέρονται για την ε, ε, ανθρωπιστική ανάπτυξη στις χώρες αυτές, ε, τις πιο φτωχές, αλλά στο να αυξήσουν τα κέρδη τους, είτε πρόκειται για την Αφρική ή για την Καραϊβική. Τώρα υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός από διεθνικές επιχειρήσεις και παραδείγματος χάρη την Κίνα και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς αυτό μπορεί ε, να βοηθήσει τις ε, ε, εκατοντάδες χιλιάδων ατόμων που θέλουν να επιλύσουν το πρόβλημα της φτώχειας μέσω του γύρου του ΠΟΕ. Και όσον αφορά τις πιστώσεις αναφέρεται εδώ ότι οι υποανάπτυξη χώρες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις και τα μία ε, προσπαθούν αλλά η κακή εμπειρία των φτωχών χωρών ακόμη και από τη δεκαετία του 1990 έχει δείξει ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σαν ένα εργαλείο για να ανοίξουν αυτές οι αγορές και αυτές οι κοινωνίες σε επιθετικές μεθόδους εισόδου και είδαμε ότι το αποτέλεσμα των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν ήταν εις βάρος των φτωχών, των μικρών παραγωγών δηλαδή οι πιστώσεις οι οποία συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις δεν είναι είναι προς όφελος ε, των ε, φτωχών ή υπέρ της ε, στρατηγικής συνοχής. Ε, υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο πριν δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή στον κύριο Ολιβιέ Μποντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η υπερ της στρατηγικης συνοχης υπαρχει καποιο αλλο σχολιο πριν δωσουμε το λογο στην επιτροπη στον πρώτα απ' όλα Χαίρετε πολύ διότι στην έκθεση αυτή λέγεται ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια θέματα. Το Συμβούλιο το συζήτησε το όλο θέμα. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζει γνωμοδότηση επί αυτού του θέματος. Τα διάφορα σημεία τα οποίοι αναφέρονται εδώ θα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, κυρίως όσον αφορά τις ε, σωστές ε, συνθήκες εργασίες, Και το θέμα της ε, ασφάλειας των ειδών διατροφής επίσης είναι σημαντικό θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι προς αυτή την κατεύθυνση προοδεύει η Επιτροπή και προσπαθεί να κάνει στον εμπορικό τομέα συνεκτικές όλες τις ε, πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειες. Σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο προσπαθούμε να έχουμε καλή συνεργασία και θα θέλαμε για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα να υπάρξει και πολιτική κινητοποίηση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πριν να δώσω το λόγο στην συντάξια γνωμοδότησης, ο κύριος Σάλμπα ζήτησε το λόγο. Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να υποστηρίξουμε πόσο μπορεί η εμπορική πολιτική να μας βοηθήσει σε θέματα ανεπτυξιακής βοήθειας. Γι' αυτό δεν μπορούμε από το ΕΛΚ αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σόλτς, διότι νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο προς αυτά τα οποία λέγονται εδώ. Στην κύριο Χιλ κάνει στα σημεία 1 και 2 πα, παπά, παπά, έκανα λάθος, αλλά ντάλλον λέω, πρόκειται για το επόμενο θέμα στο οποίο πρέπει να παρέμβω, λέει ο βουλευτής. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μαρία, έχει το λόγο. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρόεδρο ότι πρόκειται για γνωμοδότηση επί τη ουσία είναι υπεύθυνη η ΝΤΕΒΕ, η Επιτροπή Ανάπτυξης. Η Μαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια. Ίσως μέσω τροπολογιών θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στην ιδέα δημιουργίας θέσεων απασχόληση παρά το γεγονός ότι στο σημείο 2 αναφέρεται κάτι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να πω ότι στον ε, κείμενο το οποίο μπορούσα να κάνω, το οποίο πρέπει να είναι συνοπτικό, προσπάθησα να κάνω εγώ όσο δυνατόν πιο συνοπτική παρουσίαση στο σημείο τα οποία πιστεύω εγώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Όσον αφορά στην ε, χορήγηση των πιστώσεων επιμένω διότι όντως λόγω της οικονομικής κρίσης οι δυνατότητες χορήγησης πιστώσεων μειώθηκαν. Πράγμα το οποίο θα ήθελαμε να αποκατασταθεί δεδομένου ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα ε, η συνεκτικότητα μεταξύ όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πολλές φορές υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ αναπτυξιακή και εμπορικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου. Έγκριση Τη έκθεση αυτής από την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης 23 Φεβρουαρίου. Περνούμε στο σημείο 7 τη ημερήσια διάταξης. Πρόκειται πάλι για γνωμοδότηση, επειδή τη ουσία είναι υπεύθυνη η Επιτροπή ΔΕΒ, Επιτροπή Ανάπτυξης, συντάκτης γνωμοδότησης Τζο Higgins από την ΓΚΟΕ. Το θέμα είναι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής ευρωπαϊκής και η έννοια επίσημη βοήθεια για ανάπτυξη. Δίδω το λόγο στον εισηγητή, στον συντάξη, τον Τζο Higgins. Δεν θα κλείσεστε που το ΕΛΚ προσπαθεί να επιβάλλει εδώ τα αντίπεινά του. Ήταν ε, σαφές ότι οι απόψεις μου εδώ θα ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετες με το με το τι πιστεύει εδώ η ομάδα πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Αλλά εδώ επιχειρηματολογώ υπέρ του γεγονότο ότι δεν υπάρχει πολιτική συνενοχή στην πραγματικότητα. Ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει τι εμπορικέ συναλλαγές σε φτωχότερε χώρες βασίζεται σε λόγια για τις ευρωπαϊκές αρχές της δικαιοσύνη, του κάτους δικαίου και του ίσου ανταγωνισμού. Εάν κανείς διαβάσει το βασικό έγγραφο για την ε, διεθνή Ευρώπη που ανταγωνίζεται τον υπόλοιπο κόσμο ή στην αρένα του υπόλοιπου κόσμου, Νομίζω ότι καταλαβαίνει κανεί αμέσω ότι το πρώτο και το πρωτεύον ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ανοίξει όλο και περισσότερο αγορέ, να απελευθερώσει όλο και περισσότερο το εμπόριο, να απελευθερώσει όλο και περισσότερο τι υπηρεσίε στι φτωχότερε χώρε, ώστε οι ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ να μπορέσουν να δυσδύσουν και να χρησιμοποιήσουν τι χώρε αυτέ ω εφαλτήριο και πηγή για τα δικά του ωφέλη. Και αυτό χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τις τοπικές οικονομίες, τους μικρούς παραγωγούς και τους εργαζομένους. Το συγκεκριμένο έγγραφο η Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο σε μια από τις όχι τόσο επεκτεταμένες παραγράφους. του, έχει τον τίτλο «Κοινωνική δικαιοσύνη» και λέει ότι μπορεί να δούμε εδώ τις τρευλώσεις που μπορεί να προκαλέσει το άνοιγμα κάποιων ε, αγορών στις τοπικές οικονομίες και τους εργαζομένους, ιδίως για τους λιγότερο καλά προετοιμασμένους. Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι οι δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική, την Καραϊβική και την περιοχή του Ειρηνικού όχι απλώ έχουν προκαλέσει τρευλώσει στην τοπική αγορά, έχουν ε, προκαλέσει πραγματικέ καταστροφέ. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αντίφαση με τον εαυτό τη. Λέει ότι οι νέοι εμπορικοί εταίροι στη Μεσόγειο θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία στι ε, χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε, ιδίω στον τομέα τη βιοτεχνία. Αυτό πώ θα εξυπηρετήσει του φτωχότερου ανθρώπου, του εργαζομένου, πώς θα ανυψωθεί το βιωτικό της επίπεδο από την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών εμπορικών ε, σχέσεων. Ε, το άλλο επιχείρημα που προβάλλω είναι ότι όλη η διαδικασία απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης ε, για την οποία εμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές της συμφωνίες αυτό ήταν ακριβώς το πλαίσιο και η αιτία, του, του τεράστιου, της τεράστιας κρίσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της διεθνούς οικονομίας. Αυτό οι φτωχότεροι το πληρώνουν πολύ ακριβότερα από ότι οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω χάρη, που γνωρίζουν να μια αύξηση τιμών. Μεταξύ των προτάσεών μα Πρόεδρε, είναι να ακούσουμε τι μας λένε οι άνθρωποι στο δρόμο, η μικρή παραγωγή, οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστέ. Εκείνοι είναι αυτοί που έχουν ζήσει την πραγματικότητα των ε, ευρωπαϊκών εμπορικών σχέσεων και καταλαβαίνουν. Ε, εκεί ζουν και εργάζονται στην ε, απλή πραγματικότητα. Γνωρίζουν ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των όσων λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτών που προασπίζεται σε σχέση με τι εμπορικέ τη πολιτικέ και την πραγματικότητα. Και τα ζητήματα τη Σιγκαπούρη. Ε, όλη αυτή η ιδέα είναι ότι οι υπηρεσίε στι αναπτυσσόμενες χώρες οι πολιτικές ε, προμηθειών των κρατικών αρχών. Όλα αυτά πρέπει να ανοίξουν, να απελευθερωθούν για να περάσουμε στον ε, ελεύθερο ανταγωνισμό. Δηλαδή την παρήφθηση των ευρωπαϊκών και άλλων πολυεθνικών. Αυτό, κατά την άποψή μου, σε καμία περίπτωση δεν θα μας οδηγήσει στο να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την καταπολέμηση της ένδειας. Και τελευταία μου παρατήρηση, τελευταίες μου δύο μάλλον παρατηρήσεις, Πρόεδρε, σε σχετικά με τα εμπορικά πνευματικά δικαιώματα και την σχετική πνευματική ιδιοκτησία καθώς και τα φάρμακα είναι κάτι που θα ήθελα να το σχολιάσω. Ήθελα να ακούσω εδώ τις απόψεις των διαφορών ομάδων ε, τη Επιτροπή μα, Διότι τι γίνεται με τον τομέα της υγειονομική περίθαλψης και της πρόσβασης στα φάρμακα. Είναι δυνατόν να έχουμε εδώ την ίδια βίαιη προσέγγιση, τις ίδιες αρχές και μεθόδους των εμπορικών σχέσεων που θα υπαγορεύουν οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες στον τομέα της ιατρικής και της υγείας. Πραγματικά το δηλώνω ε, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια συμμετοχή, ούτε δυνατότητα βέτο από τέτοιες πολυεθνικές ή οποιαδήποτε, οποιαδήποτε εταιρεία στην πρόσβαση των φτωχότερων στα φάρμακα και την υγεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων, ο κύριος ε, Σαλβά. Τώρα, τώρα. Θα κάνω την παρατήρησή μου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κύριος Χίκκινς γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις θέσεις μας. Όπως έλεγα και εγώ, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να τονίσει ε, την ε, σημασία της ε, εξωτερικού εμπορίου για την, μεταξύ άλλων, για την βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε κάποιες παρατηρήσεις που υπάρχουν στην έκθεση της, διότι εδώ υπάρχει αντίφαση με άλλες εκθέσεις τις οποίες έχει υπερψηφίσει και ακόμη και στην Ολομέλεια η Επιτροπή μας. Στα συμπεράσματα 1 και 2 ο κύριος Χίγκινς επικρίνει σκληρά τις γενικές γραμμές της εξωτερικής εμπορικής ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγει ότι η νεοφιλελεύθερη ατζέντα της, ε, ελε, της ελευθέρωσης του εμπορίου που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια και εφαρμοστεί κατά κόρον οδήγησε ακόμη μεγαλύτερο χάρη μεταξύ πλουσίων και φτωχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ψευδές, διότι Πρέπει να πω ότι οι χώρες οι οποίες άνοιξαν τα σύνορά τους είναι χώρες οι οποίες έχουν ε, τα τελευταία χρόνια αυξήσει πάρα πολύ την ε, οικονομική τους, ε, βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση και έχουμε δει πόσο έχουν οι οικονομίες τους ωφεληθεί. Πάρτε επίσης υπόψη σας χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία και δείτε τι συμβαίνει σε κάποιες από τις δικές μας χώρες όπου η ανεργία όπως στη χώρα μου έχει φτάσει σχεδόν το 20%. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να καλέσετε την Επιτροπή να, να γνωμοδοτήσει επί της σημείο 4 γίνεται λόγος για τις ε, ΣΟΕΣ που είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο μέσον για τις εμπορικές συναλλαγές. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέμα. Επίσης, στο σημείο 5 για τα θέματα της Σιγκαπούρης νομίζω ότι είστε πάρα πολύ κατηγορηματικός πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι στις διάφορες διμερείς διαπραγματεύσεις πάρα πολύ χρήσιμες. Στο σημείο 6 γίνεται ε, λόγος για διάφορες ευελιξίες που ενσωματώνουν τη συμφωνία τρίψη να είναι σε θέση φάρμακα σε προσιτέ τιμέ. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη ο εισηγητή ε, τα σχόλια τα οποία έχουμε κάνει για τα διάφορα σημεία τα οποία έχει παρουσιάσει για να μπορέσει να αντικατοπτριστεί καλύτερα η άποψη όλων των μελών ε, στην έκθεσή του. Πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνοχή στην ε, κοινοτική ε, αναπτυξιακή βοήθεια και θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ αναπτυσσομένων και ανεπτυγμένων χρόνων για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε καλύτερα την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, τα πάντα πλην της χρησιμοποίησης όπλων. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω την πρωτοβουλία Aid for Trade, που είναι πάρα πολύ καλό μέσο αναπτυξιακή βοήθεια. Και να πω ότι είμαστε οι πρώτοι δωρητέ βοήθειας Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες του τρίτου κόσμου. Προφανώς μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι κάνουμε, αλλά αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί, θα πρέπει στην γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να αναφέρουμε όλα αυτά τα μέσα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή για να βελτιωθεί η αναπτυξική βοήθεια που χωρινεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης να αναφερθούν διάφορες ε, επιτυχίες που είχαμε στους γύρους συνομιλιών και να αναφέρουμε και τον τελευταίο γύρο της Δόχας. Επίσης θα πρέπει οι χώρες τις οποίες αποστέλλονται ή ε, βοήθεια να μπορούν να την χορηγούν εντός της χώρας τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Προφανώς εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων και τώρα ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρίσκομαι στη μέση εδώ σε σχέση με τον εισηγητή και τον προηγούμενο ομιλητή που δεν του άλλαξε ούτε το πνεύμα ούτε το περιεχόμενο της έκθεσης. Εμένα μου άρεσε το πνεύμα, αλλά συμφωνώ με πολλά από το περιεχόμενό της. Η ομάδα μου πιστεύει στην απελευθέρωση των αγορών, πιστεύει ότι το εμπόριο μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να μπορεί κανείς να το κάνει αυτό με έναν τρόπο μετρημένο. Δηλαδή δεν θέλουμε την πλήρη απελευθέρωση των αγορών. Η άποψή μου είναι επικριτική λόγω χάρη στην παράγραφο 2 του κυρίου Χίγκιν στην πρώτη πρόταση. Δηλαδή, αν ξέραμε ποια είναι η πραγματική ατζέντα που αναφέρεται εκεί για τις εμπορικές σχέσεις, θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον κύριο Χίγκιν, αλλά δεν την γνωρίζουμε. Να πω λοιπόν ότι η απελευθέρωση, το άνοιγμα μιας αγοράς δεν είναι αυτό καθ' αυτό συνώνυμο της ε, κοινωνικής πρόοδου πρέπει η ανάπτυξη να αποτελεί στόχο μαζί με την οικονομική ενίσχυση. Αλλά θα πρέπει και οι αναπτυσσόμενες χώρες να γνωρίζουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του δίνονται. Λόγω χάρη υποδομέ. Το άνοιγμα τη αγορά μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των υποδομών, αν όμω έχουν τον κατάλληλο ιστό από πριν οι αναπτυσσόμενε χώρε, μπορεί να εκμεταλλευτούν το επιπλέον δυναμικό που του δίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα το παρακολουθούσαμε. Και για τι δημόσιε προμήθειε. Εγώ δεν είμαι εχθρικό στην ιδέα οι δημόσιε προμήθειε να ανοίξουν ώστε να περάσουν ε, σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων διαγωνισμών όλοι οι παράγοντες της αγοράς. Όμως θα πρέπει να εξετάζει την νομική ικανότητα λόγω χάρη μιας αναπτυσσόμενης χώρες, χώρας να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες και βεβαίω να αποφύγουν μια ενδεχόμενη καταστροφή. Θα πρέπει όμω να υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί, οι δικηγόροι που θα γνωρίζουν και θα εφαρμόζουν του κανόνε προκειμένου να ανοίξει μια τέτοια αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι ανάλογε προποθέσει για να λειτουργήσει εύρυθμα μια τέτοια διαδικασία. Σίγουρα χρειάζεται η σωστή οικονομική και κοινωνική πολιτική των προτέρων, προκειμένου να γίνουμε τρόπο μαλό το άνοιγμα της αγοράς. Και άλλες πολιτικές νομίζω συμβάλλουν στο να δυσκολεύουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγου χάρη. Λέμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θέλουμε να φύγουν από τη θέση των απλών παραγωγών πρώτων υλών, και το είδαμε αυτό να συμβαίνει, κάποιες αγορές να ανεβαίνουν κατηγορία και να πουλούν ε, προϊόντα βιοτεχνίας ε, και τελικά προϊόντα. Και αυτό είναι σίγουρα σημαντικό. Πρέπει οι αναπτυσσόμενες χώρες να αφήσουν πλέον την παραγωγή πρώτων υλών και μόνο και να δούμε πώς λειτουργεί ως προς και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω ο κύριο Χιγκίν λέει ότι αν συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συμφωνίε ελεύθερα εμπορία με τι αναπτυσσόμενε χώρε, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και ανεξάρτητου ελεκτέ για να αποτιμούν μετά από κάποια χρόνια τον αντίκτυπο του ανοίγματο των αγορών στι τοπικέ οικονομίε. Το κάναμε αυτό. Έχουμε ήδη αποστέλει επιτροπέ ελέγχου σε διάφορε χώρε, μπορούμε να είμαστε απλώ πιο αυστηροί και πιο συστηματικοί. Θα μπορούσαμε εδώ τώρα να έχουμε έναν πολύ μακρύ διάλογο για το αν το άνοιγμα τη αγορά είναι ωφέλιμο ή όχι. Αλλά το βασικό ερώτημα νομίζω είναι αν το άνοιγμα τη αγορά συμβαίνει σε μια ήδη ανεπτυγμένη χώρα ή όχι. Τουλάχιστον επαρκώ έτοιμη γι' αυτό ή όχι. Για το TRIPS νομίζω ότι δεν έχει πολύ δίκιο ο κ. Χιγκίν. Ο μηχανισμό του TRIPS όπω έχει συμφωνηθεί επιτρέπει στι αναπτυσσόμενε χώρε να εξαιρούνται αυτού του μηχανισμού και να έχουν πρόσβαση σε φτηνά γενώσιμα φάρμακα. Εάν αληθεύουν κάποιες από τις ιστορίες μας ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ε, υπάρχει η φήμη ότι κάποιες φαρμακοβιομηχανίες ε, ενώνται να παράγουν φθηνά φάρμακα για την Αφρική λόγω χάρη. Αυτό το βρίσκω και εγώ απαράδεκτο. Θα συμφωνήσω. Και ε, σε σχέση με την έκθεση δεν μπορώ να διαφωνήσω ότι χρειάζονται κάποιε τροπολογίε. Και σε γενικέ γραμμέ είμαι σύμφωνο με το πνεύμα αλλά όχι με το περιεχόμενο. Ευχαριστούμε. Για του πράσινου ο κύριο Γιάρντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Με συγχωρείτε που άργησα. Για το σχέδιο αυτό για την ομάδα μου να πω ότι το σχέδιο κατά την άποψή μου σωστά αναφέρει τις προκλήσεις και τις ε, αντιφάσεις της πολιτικής μας, ιδίως της εμπορικής. Το ότι δεν αναφέρονται οι στόχοι της χιλιετίας, οι πολιτικές δημόσιας υγείας, αυτά είναι προβλήματα χρόνια. Ιδίως στην νέα στρατηγική Global Europe της Ευρώπης στον κόσμο. Ίσως για να ενισχύσουμε το εύστοχο αυτού του σχεδίου έκθεση, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιε περιπτώσεις λίγο πιο συγκεκριμένε ως παραδείγματα. Ιδίω στην κοινή αλληλευτική πολιτική, όπου είδαμε προσφάτως να υπάρχουν πραγματικές αντιφάσεις μεταξύ από τη μια των ευρωπαϊκών προκλήσεων σε ζητήματα ευρωπαϊκής αλληλευτικής πολιτικής και των χωρών ΑΚΕ να μπορούν να επωφεληθούν από τα τοπικά αποθέματα, το φυσικό τους πλούτο. Επίσης θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στοιχεία για τον τρόπο κατά τον οποίο τίνει να επιλύει τις διαφορές της μετρήτους η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για τις εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Ξέρουμε ότι η επιζήμια αποτελέσματα είχε η εξαγωγή γάλακτος σε σκόνη προς ε, θηγατρικές σε τρίτες χώρες από την Ευρώπη και ξέρουμε και την συμφωνία ελεύθερη, ε, ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Νότιας Κορέας. Εκεί η Ευρώπη έχει αποσπάσει εξαιρέσεις για ζητήματα εκπομπής διοξιδίων του άνθρακα από τα οχήματα εξαίρεση από την κορεατική νομοθεσία που προσπαθεί να καταπολεμήσει τις κλιματικές αλλαγές. Όλες λοιπόν αυτές τις προκλήσεις ε, πρέπει να τις δούμε από κοινού. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, προφανείς περιπτώσεις ασυνέπειας. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το κείμενο δίνοντας πολύ πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να φανεί ότι είναι εύστοχες παρατηρήσεις που γίνονται. Θα κάνουμε λοιπόν σχετικά τροποποιήσεις και εμείς από την πλευρά μας. Ε, δεν υπάρχουν άλλοι πρόσωποι από τις πολιτικές ομάδες. Όχι, λάθος. Ο κύριος Ντάρτμοντ. Πάντοτε με γοητεύει και με συναρπάζει η προσέγγιση του κυρίου Χίγγινς. Είναι πολύ εφράδης. Όμως ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με το περιεχόμενο της έκθεσής του. Αναφέρθηκε η Ινδία από τον ε, Σενιόρ Μπίντεγκεν. Ο κύριο Μάρτιν επίση έθεσε ένα ερώτημα. Το άνοιγμα των αγορών, η άρση των εμπορικών φραγμών θα ωφελήσει τι τρίτε χώρες, τι φτωχότερε χώρες. Εγώ να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Στην Ινδία με ένα πληθυσμό περίπου ενό δις ανθρώπων, ο εισαγόμενο σοσιαλισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά οδήγησε στο, μέσα σε μια πεντηκονταετία να έχει γίνει κλειστή οικονομία η Ινδία. Αντιθέτως, αν δούμε την Βρετανική πρώην απικία του Χονγκ Κόνγκ με πληθυσμό 4 εκατομμυρίων περίπου, έχουν μια απολύτως ανοιχτή οικονομία. Στην ίδια πεντηκονταετία, από το 47 περίπου μέχρι το 97, το Χονγκ Κόνγκ παραγεί εξάγει μάλλον περισσότερο σε, όχι σε κεφαλαιοχικούς όρους σε, σε σχέση με το χονδρικό εμπόριο περισσότερο με μικτούς μάλλον όρους, πολύ περισσότερο από μια χώρα που έχει πληθυσμό εναντίς ανθρώπων. Από τότε που η, η Ινδία άρχισε να χαλαρώνει τις εμπορικούς περιορισμούς της, Τότε άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά του Γκάντι βεβαίω. Και πολύ ωραία η έκθεση μας παρουσιάστηκε, μεγάλη εφράδια και πολύ μεγάλη γοητεία βέβαια, αλλά πρέπει να πω ότι διαφωνώ απολύτως. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, να πω στον συνάδελφο ότι τον κύριο Στέρντι. Στέρντι. Ευχαριστώ τον εισηγητή και πρέπει να του πω ότι ε, θα υποβάλουμε μαζί με το ΕΛΚ 5 ε, τροπολογίες. Βλέπουμε όμως ότι από τα γενώσιμα φάρμακα περάσαμε σε άλλα θέματα. Δεν είμαι πολιτικός αξιολογητής στα θέματα του Χονγκ Κονγκ και της Ινδίας, οπότε δεν έχω πολλά να πω επ' αυτού αλλά θα σας πω ότι αν θέλετε να βοηθήσετε τις υποανάπτυξη χώρες θα πρέπει να γίνει μέσω εμπορίου και όχι τόσο μέσω βοηθείας. Ε, είναι πολύ πιο αποτελεσματικού. Δηλαδή καλύτερα να τους μάθουμε να ψαρεύουν παρά να τους δώσουμε ψάρια. Ε, όπως όμως έχει λεχθεί πολλές φορές από την αρχή από όταν ξεκίνησε η Γεωργία να συμμετέχει εις ε, την ε, ε, διεθνή εμπορική σκηνή δηλαδή από το γύρο της Ουρουγουάη, έχουμε προβλήματα και πιστεύω ότι ο καθένας θα, να, θα πρέπει να μπορεί να είναι ανεξάρτητος έναντι των υπολείπων ομολόγων του. Αλλά εμείς κατά αυτόν τον τρόπο καθυστερούμε και ε, καταστρέφουμε τις ε, δυνατότητες ε, οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρξουν σε συζητήσεις εμπορικές και θα συμφωνήσω με το Γιάνν θα υποβάλλουμε κοινέ τροπολογίες με το ΕΛΚ και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να τύχουν στήριξη. Ευχαριστώ. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Ολιβιέ Μποντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένων των συζητήσεων νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να λάβει κανείς θέση. Εγώ δεν εκφράστην υπέρ ή κατά του τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα. <clears throat> Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Η απελευθέρωση δεν είναι ο μόνος παράγων ανάπτυξης και είδαμε ότι ορισμένες χώρες οι οποίες προχωρούν ε, ε, ε, στην καταπολέμηση της στόχιας μπορούν να συγκριθούν με άλλες που δεν προχωρούν καθόλου. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου υπάρχουν επίσης δυνατότητες απελευθέρωσης, Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των υποανάπτυξης χωρών. Ε, αναφέρομαι στο γενικευμένο σύστημα των προτιμήσεων ή τις ε, ε, ε, παροχές οι οποίες δίδονται και επίσης οι πολιτικές ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη υπάρχουν ακριβώς για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη και μεταξύ των προτεραιοτήτων για να υπάρχουν συνεκτικές πολιτικές είναι η ε, διατροφική ασφάλεια και οι συμφωνίες ε, αλληλείας οι οποίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν τώρα και ελπίζω ελπίζουμε ότι ήδη θα υπάρξει μια εξέλιξη πέραν αυτής η οποία έχει ήδη σημειωθεί. Δηλαδή τώρα υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ε, για τη χορήγηση δημοσιονομικών ε, ε, ενισχύσεων δηλαδή δεν αγοράζουμε μόνο δικαιώματα αλληλείας αλλά δίδουμε και ενισχύσεις οι οποίες συνδυάζονται με ορισμένες προϋποθέσεις για να υπάρχει πιο συνεκτική αντιμετώπιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η συνάδελφός μου που κάθε δίπλα μου έδειξε ότι ορισμένα θέματα ήταν απλούστατα παροδικά, διήρκεσαν έξι μήνες. Μπορεί κανείς να σχολιάσει την σκοπιμότητά τους, αλλά υπήρξαν ορισμένες πολιτικές επιλογές που απέδωσαν ή όχι. πιστεύω ότι η νέα προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πολιτική αναπτύξεως πρέπει να εστιαστεί εις την διατροφική ασφάλεια, στις κλιματολογικές αλλαγές, στις μετακινήσεις πληθυσμού, την ασφάλεια και το εμπόριο βέβαια και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι πολιτικές ε, δια αλληλεπιδράσεως Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την ε, νέα μορφή η οποία θα προέλθει από αυτές τις προτάσεις και όσον αφορά τους αριθμούς οι οποίοι έχουν υποβληθεί πιστεύω ότι η μείωση η οποία ε, έχει δοθεί στο Aid for Trade ε, συνδυάζεται με μειώσεις διότι είναι ένα εργαλείο κατόπιν ετήσεως όταν δηλαδή έχουν οριμάσει τα προγράμματα και πρόκειται για προγράμματα υποδομής δηλαδή ένα χρόνο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ε, και την επόμενη χώρα τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχουν έτοιμα όριμα προγράμματα και γι' αυτό μειώνουν τις στατιστικές κάπως έτσι πρέπει να αξιολογηθούν Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο και πάλι στον εισηγητή για να αντιδράσει όσον αφορά τα σχόλια Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένος ότι ε, η ευλωτία μου επηρέασε τον ε, Λόρδο Ντάρτμουρ τον οποίο μπορώ να προσφωνήσω ως Σαρλ βεβαίως ε, σκεφτείτε τι θα γινόταν πριν από 200 χρόνια. Ε, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε το πρότυπο της δημοκρατικής ε, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στον κόσμο αλλά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας η τάξη σας μας χορήγησε το δικαίωμα ψήφου μετά από σκληρούς αγώνες. Βεβαίως ε, δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Ζάλμπα και οι χριστιανοδημοκράτες ε, θα αντιταχθούν ε, σκληρά στα θέματα τα οποία έχω υποβάλει διότι ε, υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Οι χριστιανοδημοκράτες, το ΕΛΚ είναι αυτοί οι οποίοι προώθησαν ε, την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση τα τελευταία 20 ε, χρόνια και μας οδήγησαν στην κατάσταση που έχουμε σήμερα. Εάν λοιπόν θέλετε τα ίδια που κάνετε στην Ευρώπη να τα κάνετε και σε άλλες χώρες, διαφέρουν ουσιαστικά οι απόψεις μας ε, θα υπάρξουν οι τροπολογίες φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία παρουσίασα θα έχει αλλάξει όταν ε, θα, βάλουν το χέρι τους ε, οι άλλες πολιτικές ομάδες αλλά παρουσίασα απόψεις που πιστεύω αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων στις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ε, συνάψει εμπορικές ε, σχέσεις. Ο κύριος Στέρντι είπε ότι είχαν συζητηθεί διάφορα θέματα, τα φάρμακα, τα τρόφιμα και αυτό δεν είναι περίεργο διότι όντως ο εμπορικός μηχανισμός είναι πολύπλευρος. Όσον αφορά τον κύριο Σάλβα δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε απλώς σε τρεις χώρες, δηλαδή την Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα, που είναι ένα παράδειγμα του ανεπτυγμένου εμπορίου, αλλά είναι πολύ επιλεκτικός, διότι επέλεξε τις πιο ισχυρές χώρες και αυτές μπορούν όντως να κινηθούν ανεξάρτητα ε, να αντιθέσει με τις πιο αδύναμες και τις πιο μικρές οικονομίες οι οποίες ε, ε, δεν σημαίνουν ότι δεν συμφωνώ ότι ε, ότι συμφωνώ ότι η ε, ζωή για τους εργαζόμενους είναι παράδεισος. Ή στην Κίνα και στη Βραζιλία υπάρχει μεγάλη καταπίεση των εργαζομένων. Έχετε ακούσει την κοινωνία των πολιτών, το, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, τι κακό έχει κάνει περιβαλλοντολογικά η ανάπτυξη στη Βραζιλία ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τι λένε ε, ε, οι άνθρωποι, ο απλός λαός που ζει στις διάφορες περιοχές. Αντί να γενικεύουμε και να προσποιούμαστε ότι δημοκρατικές ευρωπαϊκές αρχές και η ερμηνεία που δίνουν στο εμπόριο είναι οι ίδιες με αυτές τις οποίες ακούν και καταλαβαίνουν και οι απλοί άνθρωποι επιτόπου. Ε, φαντάζομαι ότι οι πολιτικές ομάδες θα επανέλθουν και εγώ θα επανέλθω με ε, παραδείγματα για να αποδείξω ότι τα ε, θέματα τα οποία φύγω έχουν κραυγαλαία παραδείγματα τα οποία τα στηρίζουν. Ευχαριστώ. Προς ενημέρωση η ε, λήξη ε, ε, της προθεσμίας είναι 2 Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες και παρόλες τις διαφορές απόψεων που έχουμε ελπίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια ισχυρή γνωμοδότηση η οποία θα στηριχτεί από την πλειοψηφία. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 8, ανταλλαγή απόψεων με ε, τον ε, πρέσβη Ρικάργο Νεβερταβάρης που είναι ήδη εδώ για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ρεζιλίας. Ε, υπομορφήν ε, εισαγωγής θα ήθελα να πω ότι προτού δώσω τον λόγο των ε, καλεσμένων μας το δημογραφικό βάρος της Βραζιλίας στο πρόσφατο παρελθόν ε, ε, την, καθιστά ε, τον ηγέτη στην Νότιο Αμερική, στη Λατινική Αμερική και καλύπτει το 1 τρίτο του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αυτή την περιοχή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή ε, υπήρχαν ε, 27 ε, εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ενώσεως που αυξήθηκαν κατά 65% ενώ διπλασιάστηκαν και οι εισαγωγές. Ε, Ζητείται μία συμφωνία ελευθέρων εμπορίου με το Mercosur ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών του Μερκοσούρ και να υπάρχει απελευθέρωση του εμπορίου και των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών συνόλων ομάδων διότι είχαμε σημαντικές ε, ε, ε, σημαντικές συναλλαγές ε, από το 2000 ε, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις οι οποίες σταμάτησαν το 2004 διότι και οι δύο πλευρές περιμένουν ε, την ευτυχή έκβαση του γύρου της Ντόχα και δεδομένων των δεσμεύσεων των χωρών και ε, της ε, σημασία του για την παγκόσμιο ε, οικονομία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Βραζιλία είναι σημαντικός εταίρος στο διεθνές εμπορικό σύστημα και γι' αυτό την επόμενη άνοιξη θα επισκεφθεί μία αντιπροσωπεία μας στη Βραζιλία και θεωρούμε ότι αυτή η ε, επίσκεψη θα είναι πολύ σημαντική για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας ε, και τις σχέσεις μας με τη Βραζιλία όσον αφορά και το γύρο της Ντόχα και τις εμπορικές και τις οικονομικές σχέσεις. Με τα πολύ μεγάλης χαράς λοιπόν χαιρετίζω τον πρέσβη Ρικάρντο Νέιβα Ταβάρες ο οποίος είναι επικεφαλής αποστολής της Βραζιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και με τα μεγάλης χαράς θα σας ακούσουμε. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει ε, τη συζήτηση αυτού του θέματος στι 11.30. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρά το γεγονό ότι εσείς μιλήσατε αγγλικά, κάτι το οποίο πάντα με ενθουσιάζει όταν είμαι στο κοινοβούλιο είναι ότι έχω πάντα την δυνατότητα να μιλήσω πορτογαλικά. Με την ε, ε, βραζιλιάνικη προφορά με βέβαια, αλλά θα μιλήσω λοιπόν πορτογαλικά. Κύριε Βιτάλ Μορέιρα, πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότικα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, Διεθνούς Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που με απευθύνατε να λάβω το λόγο στην Επιτροπή σας και να κάνουμε αντάλογη απόψεων για το θέμα της σημερινής συγκυρίας όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις Βραζιλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσδίδω ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συνάντηση δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει όλο και πιο σημαντική θέση στην εξέλιξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας. από τον προηγούμενο Δεκέμβριο ξέρουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας που ενισχύει και το λόγο, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε σε μια παράδοξη συγκυρία σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε τις παγκόσμιες οικονομίες από το τέλος του 2008 πρέπει να πω ότι δημιούργησε ε, μεγάλο προστατευτισμό στον περισσότερο κόσμο. Ευτυχώς, χάρη στις διάφορες ε, εμπορικές πολυμερείς συμφωνίες μπορέσαμε να αντισταθούμε σε αυτή την διαδικασία. Απ' την άλλη πρέπει να πω ότι στην, κατά την ε, διάρκεια αυτής της ε, κρίσης είδαμε ότι οι κατεβλήθησαν συγκεκριμένες και μεγαλύτερες προσπάθειες από όλες τις κοινωνίες για να μπορέσει να βελτιωθεί το διεθνές εμπόριο. Και πρέπει να πω ότι διάφορες επιχειρήσεις μπόρεσαν να επιπλέψουν. Είναι λοιπόν στα πλαίσια αυτής της ε, συγκυρίας πολύ σημαντικό να μπορέσει να υπάρχει ε, ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα για να μπορέσουν να περιχαραχωθούν οι διάφορες πολιτικές ε, ε, προστατευτισμού και να μπορέσουν οι διάφορες εμπορικές συναλλαγές να βελτιωθούν. Πρόκειται για γύρο ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια ισχύει και ακόμη δεν έχει μπορέσει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να ληφθούν υπόψη πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών. Γι' αυτό ε, πρώτα απ' όλα υπάρχει εδώ το θέμα της ε, ε, λήψης υπόψη των διάφορων συμφερόντων των απτυσσομένων χωρών. Ποιος ε, θα μπορούσε να φανταστεί στην αρχή ότι η συμμαχία μεταξύ το, ε, περίπου 20 αναπτυσσομένων χωρών θα μπορούσαν να αντισταθούν στις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις. Με μεγάλη λοιπόν ευχαρίστηση. Εμείς στην Βρασιλία διαπιστώνουμε ότι με αυτή την ε, συμμαχία στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα ε, ενισχύθηκαν οι θέσεις μας και σήμερα καταλήξαμε να έχουμε περισσότερες συγκλίνουσες απόψεις παρά αποκλίνουσες διάφορα θέματα ώστε να υπάρχει ε, στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής λυσμένη άποψη για τα διάφορα εμπορικά θέματα. Πρέπει να πω ότι εμείς ε, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε το 2010 να ολοκληρώσουμε το γύρο της Δόχα έτσι όπως αποφασίστηκε πέρσι στην ε, διάσκεψη υπουργών στο Δελχείο. Κύριοι και κύριοι βουλευτές, οι εμπορικέ σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωσης Βραζιλία πρέπει να πω ότι αναπτύχθηκαν τα 10 τελευταία χρόνια. Από το 1998 έως το 2008 αυξήθηκαν οι εξαγωγές κατά 56% προς την Βραζιλία. Όντως το 2009 υπήρξε μία μικρή στασιμότητα, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Βλέπουμε όμως τώρα σημεία ανάπαξης. Από την πλευρά τώρα της Βραζιλίας, οι διμερείς ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι θετική, πρέπει να πω ότι είναι και ποιοτική η εξέλιξη. Το παρελθόν οι δικές μας εξαγωγές χαρακτηρίζονταν από υπερίσχυση βασικών προϊόντων. Σήμερα βλέπουμε όμως ότι περισσότερο από τις μισές μας εξαγωγές προϊόντων πρόκειται για επεξεργασμένα προϊόντα. Πρέπει να πω ότι οι προϊόντα τα οποία εξάγουμε είναι ε, σόγια, καφέ, ε, καύσιμα, αλλά επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε και εξαγωγή ε, τεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων αεροσκαφών, ε, αυτοκινήτων και τα Η, στον τομέα των μεταφορών της ηλεκτρικής ενέργειας και των ε, μηχανικάτων, πρέπει, μηχανημάτων πρέπει να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλές ε, εξαγωγές. Σας είπα ότι έχουμε ποιοτική ξέλιξη των συναλλαγών μας στο παρελθόν ε, η σχέση μεταξύ μας ήταν ασυμμετρική και είχαμε κυρίως ε, ροή αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη, προς Βραζιλία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο ισοσκελισμένα. Το 2008 έγιναν επίσης και μεγάλες επενδύσεις ευρωπαϊκές προς την Βραζιλία. Το 2008 οι επενδύσεις οι κοινοτικές ήταν 22,5 δις και οι δικές μας επενδύσεις ήταν επίσης περίπου οι ίδιες. Τα ο... Φέλη είναι αμοιβαία και φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. 2005 στα πλαίσια της Μερκοσούρ προσπαθήσαμε ε, να προσεγγίσουμε περισσότερες διάφορες χώρες. Δεν θα σας πω τώρα ποιες ήταν οι λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι δύο εταίροι ε, μπόρεσαν να γεφυρώσουν το μεγάλο χάσμα που υπήρχε μεταξύ τους από το 2004. Σήμερα κατά την εκτίμησή μας υπάρχει ε, δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και οι περισσότερες δυσκολίες προέρχονταν από το ότι μαζί με τις συζητήσεις στα πλαίσια του Μέρκοσουρ γίνονταν και οι διάφορες συζητήσεις στα πρέσια του γύρου της Δόχα. Σήμερα ε, προσπαθούμε να συντονίσουμε καλύτερα τι προθέσει μα και ξέροντα ποιε είναι οι δυνατότητε των μέχρι των ΔΕ, καταβάλουμε προσπάθειε ώστε να μπορέσουν οι διάφορε περιφερειακέ διαπραγματεύσει που κάνουμε να ολοκληρωθούν με επιτυχία. Στο τέλο του 2008 πρέπει να πω ότι κατέβαλε μεγάλε προσπάθειε η Βραζιλία ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να επωφεληθεί από τις ε, δυνατότητες που προσφέρονται και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε καταρχάς στις διάφορες ερευνητικές συναντήσεις που έγιναν πέρσι. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα γιατί σήμερα η οικονομική κατάσταση δεν είναι ανθυρή. Ξέρουμε ποιες είναι οι περισσότερες ε, δυσκολίες αλλά για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η διαπραγμάτευση θα πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και όχι τι είναι ιδεατό. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την θέση των Ευρωπαίων να ε, κάνουν διάφορους περιορισμούς στο θέμα των αγροτικό πράγμα, το τομέα τον οποίο ε, για τον οποίο εμείς έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει λοιπόν με πνεύμα κατανόησης και ευαισθησίας να αντιμετωπίσουμε τι διαπραγματεύσει σε αυτό το τομέα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επίση στον τομέα των υπηρεσιών και τη βιομηχανία. Πιστεύω ότι ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει ε, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και με την κοινή λογική. Αυτό το οποίο λέγουν common sense ε, οι αγγλόφωνοι. Πιστεύω λοιπόν ότι με τέτοιο πνεύμα λογικής θα πρέπει να δούμε τις ε, σχέσεις εμπορίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ε, βοηθήσει να βελτιώσουμε τις εμπορικές μας ε, σχέσεις. Ε, το ότι είμαστε από το 2007 και μετά στρατηγικός εμπορικός εταίρος είναι κάτι το οποίο μας βοηθά και εμάς και εσάς και κυρίως αποδεικνύει ότι υπάρχουν, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των ε, σχέσεων και της, του ωφέλους, του αμοιβαίου του οποίου μπορεί να αποτελέσουν αυτές οι συναλλαγές και για μας και για σας. Υπάρχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον και βεβαίως όσο περισσότερο ε, αυξάνουν και διάφορες εμπορικές ροές τόσο περισσότερο θα πρέπει να γίνουν διάφορες προσαρμογές ε, δεδομένου ότι θα θέλουμε να καταλήξουμε σε πάρα πολύ ε, καλό επίπεδο ανταλλαγών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκλησή σας. Πρέπει να σας πω ότι ζούμε αυτή τη στιγμή μία περίοδο μεγάλων αλλαγών. Η ταχύτητα των οποίων μας κάνει να λέμε ότι στον γης μέλλον ο κόσμος δεν θα μοιάζει με αυτόν που ξέρουμε σήμερα. Η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να υποφεληθούμε θετικά από αυτές τις αλλαγέ χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε σε μέσα που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν. Η Βραζιλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει το ρόλο της στον εμπορικό τομέα και γενικότερα στην διεθνή σκηνή δεδομένου ότι ο προστατευτισμός τον οποίο δεν επιθυμούμε εμείς είναι απλώς μια απόπειρα να παραμείνουμε στα παλαιά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Χαϊδεύει τα αυτιά μας αυτή η εξαιρετική βραζιλιάνικη προφορά σας, κυρίως εμένα ως Πορτογάλο. Θα ήθελα να σας πω προσωπικά Χαίρομαι και είμαι υπερήφανος που είμαι Ευρωπαίος, αλλά έχω και κάποιες ρίζες στην Πορτογαλία. Έχω και οικογένεια στην Πορτογαλία, άρα αντιμάχονται τα συμφέροντα μέσα μου. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να λάβουν μέρος στην συζήτηση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε στη διάθεσή μας 20 λεπτά. Ο κύριος Αρεύσκη. Αριστερά μου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρέσβη για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Βραζιλίας, οικονομικές σχέσεις. Αυτές οι δυνατότητες τις οποίες και αγραφήσατε είναι πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αναφέρεται στο συντονισμό της ε, εμπορικής πολιτικής από πλευράς της Βραζιλίας με άλλες χώρες από το, την ομάδα BRIC, δηλαδή ε, ε, Βραζιλία, ε, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Θα ήθελα να ξέρω τι συντονισμός υπάρχει μεταξύ των χωρών αυτών. Οι χώρες BRIC έχουν μία ενιαία θέση προς τον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερη ερώτηση. Πώς ε, αναμένετε την ε, βραζιλιανή οικονομία να εξελιχθεί στο μέλλον όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε κάποια νέα τάση όσον αφορά την, την ε, βιομηχανία της Βραζιλίας, της τάσης στον τομέα της οικολογίας. Δηλαδή ε, στο μέλλον θα μπορεί η Βραζιλία να προσφέρει μοναδικές λύσεις και να αποτελέσει ένα πιο ενδιαφέροντα ομόλογο ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο στον κύριο Μενέντες και τον παρακαλώ να περιοριστεί σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη πριν να κάνω τις συγκεκρισμένες παρατηρήσεις ως σοσιαλιστής, πανώς θα ήθελα να συγχαρώ τη Βραζιλία για την ενεργητικά μετριοπαθή του θέση που έχει στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο στα πλαίσια των χωρών της Λατινικής Αμερικής, αλλά κυρίως στη σχέση με τις χώρες ε, τις αραβικές. Και τώρα θα ήθελα ε, να κάνω τις παρατηρήσεις μου. Μας δώσατε εσείς κύριε Πρόεδρε κάποια στοιχεία. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω στη σημασία των σχέσεών μας. Απλώς θα ήθελα να ότι Όλοι θέλουμε να προχωρήσει ο γύρος των συνομιλιών στην Τόχα. Και θα πρέπει να καταβάλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για να συμβεί αυτό. Όχι μόνο για να μπορέσει να υπάρξει τελικά συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας, αλλά μέσω της, των συνομιλιών του γύρου της Δόχας να μπορέσει να αμβληνθεί η φτώχεια στις χώρες Λατινικής Αμερικής ε, γενικότερα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον ε, πρέσβη της Βραζιλίας. Θα ήθελα η στρατηγική λύση την οποία υποστηρίζουμε να χρησιμεύσει για να επιληθούν κάποια προβλήματα ε, στο τομέα των επικοινωνιών, των υπηρεσιών, την πρόσβαση κάποιων ευρωπαϊκών εταιριών στα δημόσια έργα, την προστασία ε, την... Ε, παραποίηση, πολέμηση της πειρατείας και άλλα θέματα. Ως ε, Ευρωβουλευτής πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι όλοι θέλουμε οι σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο με τη Βραζιλία να είναι επιτυχής. Είναι προφανές ότι όπως είπε ο κύριος πρέσβης από το 2004 δεν έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Μερκοσούρ. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πει και να ψήσει του κύριο Πρέβη ποιε είναι τα κύρια, η, η, πρόοδο στην οποία μπορούμε να περιμένουμε στο γύρο της Δόχα, καθώς και στο θέμα της ε, επανάληψης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες Μερκοσούρ σε σχέση με την διάσκεψη κορυφής που θα κάνουμε με τις χώρες Καραβικής το ε, Μάιο στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Κύριο Στέρντι, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον ε, πρέσβη για την ε, συζήτηση αυτή που έχουμε μαζί. Ήθελα να σταθώ σε ένα-δυο ζητήματα στα οποία μπορεί και να μην απαντήσει λόγω τη διπλωματική του θέση, ιδίω το πρώτο, αλλά θέλω να το θέσω ούτω ή άλλω το ερώτημα. Στο γύρο τη Ντόχα ξεκινάμε με μια κατάσταση που μα υποχρεώνει να φέρουμε τι ΗΠΑ στο τραπέζι αλλιώ των συζητήσεων. αλλιώ δεν θα υπάρξουν πραγματικά διαπραγματεύσει. Τι θα κάνει η Μερκοσούρ για να μα διευκολύνει. Το λέω αυτό και όλα στο πλαίσιο και ίσω αυτό να μην σα αρέσει, ότι η οικονομική κρίση με το δάνειο τη Αργεντινή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει εντός της, ε, του, της ομάδας Μερκοσούρ. Πολλοί βουλευτές και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ ε, αναρωτιούνται αν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Για τη βιοεθανόλη τώρα. Ένα από τα βασικά σας εξαγωγικά προϊόντα και πάλι ασκούνται πιέσεις προς τους ε, βουλευτές γενικώ και το Κοινοβούλιο από τους εκλογείς του για την βιώσιμη και την καλλιεργήσιμη ε, γη και τις πρακτικές που μπορεί να εφαρμόζονται στη γη αυτή. Ε, λαμβάνουμε πολλές ε, επιστολές σχετικά. Μπορείτε να μας αβεβαιώσετε ότι τα τροπικά δάση της Βραζιλίας δεν θα καταστραφούν περαιτέρω για την καλλιέργεια ε, των, ε, της <clears throat> και για τη σόγια, για τα προϊόντα σόγιας, πρέπει να πω ότι είμαι υπέρ των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Είναι τεράστια ευκαιρία να εξεύρουμε τρόφιμα για τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως όταν υπάρχει έλλειμμα. Ποια είναι η κατάσταση και άποψή σας σχετικά. Uh, Επειδή έχουμε και χρονικούς περιορισμούς, νομίζω να περιοριστούμε αυστηρός σε δύο λεπτά για την κάθε παρέμβαση. Ο κύριος Φέλνερ. Τρία σόκερ. Eh, först och främst eh, direktinvesteringar. Κύριε Πρέσβη, ήθελα να θέσω και εγώ... Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στην παραγωγή και στη διαφοροποίηση ε, του εμπορίου. Μιλήσατε ε, για τη διαφοροποίηση ε, του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία μονομερής αντιμετώπιση ίσως λόγω της οικονομικής κρίσης. Εκπροσωπώ τη Σουηδία εδώ που είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη Βραζιλία και ελπίζω ότι και μετά την οικονομική κρίση θα συνεχίσει να είναι μεγάλος επενδυτής ε, ε, η Βραζιλία και οι επενδύσεις είναι ένα βασικό θέμα της ε, εμπορικής συνεργασίας Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν οι σχέσεις ώστε να υπάρχει κάποια προτεραιότητα για τις εμπορικές επενδύσεις. Όσον αφορά τις εξαγωγές, μ' αρέσει και ο καφές και το βοδινό κρέας. Τι γίνεται όμως με τις διαμάχες, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τις συναλλαγές αυτών των γεωργικών γεωργικών προϊόντων χωρίς να συμβάλλουμε στα εμπορικά εμπόδια και μιλήσατε για διαφοροποίηση των γεωργικής παραγωγής. Μπορεί να κάνει κάτι η Ευρώπη να σας βοηθήσει από αυτό για να επωφεληθούμε όλοι και εμείς στην Ευρώπη και εσείς. Ευχαριστούμε. Και κύριος Ράντο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγχαρητήρια και για τι απαντήσει αυτέ που δώσατε στον πρέσβη. Το βρίσκω πολύ πιο σύγχρονο τρόπο προσέγγιση από το φάσμα της ε, νέα απεικιοκρατία. Πρέπει να πω ότι εγώ εκτίμησα ιδιαίτερα την παρέμβαση του κυρίου Λούλα στην Κοπενχάγη. Ήταν στο ύψο των προκλήσεων των σημερινών και δεν παρενέβη για να πει τι δεν κάνουν οι άλλοι, αλλά τι είναι έτοιμη να κάνει η ίδια η Βραζιλία. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτή την άποψη το παράδειγμα αυτό πρέπει να ακολουθηθεί και να βρει μιμητέ. Τώρα, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών κατά πρώτον. Η Βραζιλία πώ σκέφτεται να χρησιμοποιήσει εμπορικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη πέραν τη μεταφορά τεχνολογιών, τη μεταφορά περιβαλλοντικών αγαθών για να καταπολεμήσει ακριβώ τι κλιματικέ αλλαγέ. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Η αποψήλωση των δασών. Κατά πρώτον, ισχυρό παράγοντα για να δούμε αν θα καταπολεμηθούν κλιματικέ αλλαγέ ή όχι. Η Βραζιλία λοιπόν επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυστηρότερα τα μέτρα τη για την παράνομη αποψήλωση, την υλοτομία και θα επιτρέψουμε στις βραζιλιάνικες αρχές να εξάγουν προϊόντα που φτάνουν στην Ευρώπη χωρίς να ανταποκρίνονται στα πρότυπα για την νόμιμη εμπορία σχέση με τα κριτήρια που ισχύουν για τον τομέα αυτό. Και μετά για τα βιολογικά καύσιμα. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερως. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη των ε, καυσίμων αυτών έχει να κάνει και με ζητήματα επισητιστικής ασφάλειας, ε, φτώχειας του πληθυσμού και της αποψήλωσης των δασών θα πρέπει τα κριτήρια τα αυστηρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθούν, πιστεύετε, και να ισχύει το εμπάργκο, το μορατόριο με αυτό για, τα, για την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Βραζιλία και για τα γενώσιμα φάρμακα. Στις κάτω χώρες ε, μια παρτίδα τέτοιων φαρμάκων που κατευθυνόταν στην Βραζιλία μπλοκαρίστηκε πριν την εξαγωγή της τι ζήτηση, τι μάλλον εκκλήσεις θα αποφύγετε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην συμβαίνουν αυτά πλέον. Πρόεδρος, εγώ προσωπικά δεν έχω οικονομικά συμφέροντα στην Βραζιλία, Ομολογουμένω. Κύριε Βίνκλερ, είναι η δεύτερη φορά που ε, έχετε την ευκαιρία να παρέμβετε για 1,5 λεπτό αυτή τη φορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα παραμείνω στο περιθώριο αυτό. Θα σα ζητήσω ένα λεπτό, αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και λίγα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσω τον πρέσβη για τις ε, πολύτιμε πληροφορίε που μας έδωσε. Θα ήθελα να του θέσω ένα ερώτημα ίσω διμερό, διότι η πολυμερής διάσταση ήταν κάτι που φάνηκε και από την συζήτηση με του υπόλοιπου συναδέλφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου 11 δι ε, ευρώ εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με τις χώρες σα. Για την προστασία της αγοράς στην Βραζιλία, σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη προστασία από ό,τι θα θέλαμε ή θα επιθυμούσαμε και συζητήσαμε με τον πρέσβη για το ρυθμό με τον οποίο όλα αυτά αλλάζουν και για το τι ευκαιρίες υπάρχουν και μπορεί να διατίθενται πλέον. Μιλήσατε για την μείωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών όπως ισχύουν στη βραζιλιάνικη αγορά. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και ακόμη δύο δευτερόλεπτα για να τονίσω αυτό που ο συνάδελφος και αντιπρόεδρος είπε. Για το σχόλιο που έγινε για την πρωτοβουλία και την ομάδα BRIC. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα και άλλοι ότι είναι πραγματικά μια αυθεντική μορφή συνεργασίας. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Να πω ότι ο πατέρας μου ήταν για 20 χρόνια πρόεδρος της Αγγλοβραζιλιάνικης, του Αγγλοβραζιλιάνικου Συλλόγου και η δεύτερη σύζυγός του, η θετή μου μητέρα, ήταν Βραζιλιάνα. Βλέπουμε ότι γίνονται τεράστια άλματα στην βραζιλιάνικη οικονομία. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της κεντροαριστεράς στη Βραζιλία παρόλα αυτά δεν εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο. Θα ζητούσα λοιπόν από τον πρέσβη και τους συναδέλφους του να έχουν κατά νου και την τοποθέτηση του επικεφαλής της Βραζιλιάνικης Αντιπροσωπής παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και στενοί και προσωπικοί δεσμοί μεταξύ της Βραζιλίας και των ε, μεμονωμένων χωρών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ίσως ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται καλύτερα παρά ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε ο κύριος Higgins από την ΚΟΕ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ο συνδυασμό εμπορίου και δικαιοσύνη στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση με, με την Βραζιλία πρέπει πιστεύω να βασίζεται στη δικαιοσύνη και του πώ διαθετεί τα ζητήματα γη η Βραζιλία στο εσωτερικό τη. Όταν ο Νάσο Ντασίλβα πήρε την εξουσία, υπήρχαν ε, πολλέ ε, ε, προσδοκίες για αναδασμό μεταξύ εκατομμυρίων ε, πολιτών της Βραζιλίας, αλλά και τεράστια απογοήτευση έχει επέλθει λόγω της καθυστέρησης. Στο Σανταρέμ, λόγου χάρη, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έχουν καθόλου γη. Υπάρχουν ε, σύλλογοι γεωργών, συνδικαλιστικές οργανώσεις γεωργών που πιέζουν, πιέζουν για να μην είναι πλέον ακτήμονες. Και όταν εγώ πριν από λίγα χρόνια πιστεύτηκα το Ρίο Γκράντε του Σουλ, όχι, με συγχωρείτε, άλλο κράτο είναι, θα το θυμηθώ εντό ολίγου. Τέλο πάντων, είδα μεγάλα αγροκτήματα που καλλιεργούν σόγια και ζαχαρότευτλα και μεγάλα κοπάτια βοηδών. Ενώ σε χωριά ηθαγενών εκεί δίπλα, παιδιά πέθαναν από, πέθαναν από ε, υποσυντισμό. Τι κάνει λοιπόν ε, η Βραζιλία για να επισπεύσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έπειτα υπάρχουν και τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά που είναι πήγοντα. Η Βραζιλία έχει την ε, χαρά να έχει την, τον Αμαζόνιο στα εδάφη της, ε, τη, τα δάση του, τη ζούγκλα. Όλα αυτά είναι καθοριστική σημασία για τα οικοσυστήματα παγκοσμίω. Όμω έχουμε διαρκή παράπονα και αποδεκτικά στοιχεία από του ντόπιου σε ό,τι αφορά την αντιπεριβαλλοντική πολιτική και τις ενέργειες κάποιων βασικών ε, οργανισμών που έχουν τη βάση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν για συγκεκριμένες εταιρείε, πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες για καταστροφή του περιβάλλοντος σε περιοχές δυτικά του Ρίο Ντεζανέιρο και απειλές προς τους ντόπιου να αναχαιτήσουν αυτές τις ε, πολιτικές. Ε, Πολλέ οικογένειε οδηγούνται σε εξόντωση με τι μεθόδους αυτές. Τι θα ασχοληθεί θα ο κύριο Πρέσβης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ε, δύο θέματα που ήταν στο επίκεντρο, την ε, περιφερειακή συνεργασία και τις ε, επιπτώσεις για την, τις εμπορικές σχέσεις. Δηλαδή, ε, πώς τοποθετήσετε ε, σχετικά με τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Βραζιλίας και άλλων χωρών Λατινικής Αμερικής και δεύτερον, πώς αντιμετωπίζετε τις εμπορικές σχέσεις, διότι υπάρχουν περιφερειακές ευρωπαϊκοί συνασπισμοί. Εσείς λοιπόν τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορείτε να ενισχύσετε την συνεργασία και ποιοι παράγοντες θα σας επηρεάσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριος Άνιας δεν θέλει το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε το, λόγο να δώσουμε, το χρόνο να δώσουμε το λόγο και στην Επιτροπή. Θα έχουμε όμω άλλε ευκαιρίε στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, θα καλέσω τον προσκεκλημένο μα να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, α πούμε. Είστε πολύ γενναιόδωρο. Πρόεδρο, ε, προσπαθήστε, θα σα δώσω και μερικά λεπτά αν χρειαστεί. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είναι λίγο δύσκολο θα χρειαστώ πολύ περισσότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες αργότερα από την αντιπροσωπεία μας, εφόσον χρειαστεί. Μια επιπλέον συνεισφορά για τη συζήτησή σας σε μεταγενέστερο στάδιο. Για το ζήτημα του TRIPS, πρώτα απ' όλα. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είμαι παρόν στην πρώτη συνεδρίαση αυτή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από τη στιγμή αυτή, πριν από μερικά χρόνια και μετά, αναπτύσσουμε έναν διάλογο διαρκή και μια συνεργασία επίσης διαρκή. Διοργανώσαμε συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και εξακολουθούμε να βρίσκουμε κοινό έδαφος συνεννόησης και κοινά συμφέροντα. Αυτό δεν ξεκίνησε βέβαια από το μηδέν, διότι συντονισμό έχουμε διενεργήσει σε πολλά, διαφορετικά, σε πολλά και διάφορα πολυμερή φόρα για Πολλού από του τομεί που μα ενδιαφέρουν και στα πλαίσια των παραδοσιακών ε, σχέσεών μα με τις περισσότερες χώρες εταίρου και στα πλαίσια της συνεργασία BRIC. Έχει λοιπόν επιτελεστεί πρόοδο και αυτό θα συνεχιστεί νομίζω. Τώρα για την πρωτοβουλία για την ομάδα BRIC είναι γνωστά αυτά. Πρόσφατα στο Financial Times διάβασα μια σειρά άρθρων όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μια συνεργασία εν εξελίξη για όλους. Για την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις κοινοτόμες τεχνολογίες και ούτω καθεξής, πάρα πολλά θα είχα να πω. Ένα από αυτά είναι ότι το σύστημα που θεσπίζουμε με τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, επακριβώς προβλέπει το διάλογο για την επιστήμη και την τεχνολογία. Ο πρώτος τομέας που καλύπτεται είναι η εθανόλη. Θα το θίξω ευθύ αμέσω το θέμα τη βιοεθανόλη. Αλλά είναι ένα από τα προϊόντα αυτό το οποίο διαρκώ αναπτύσσεται στην Βραζιλία τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Και έχει αποδείξει την επιτυχία του καθώς ακόμη και τα μοτίβα κατανάλωσης ε, ενέργειας στη χώρα μας έχουν μεταβληθεί εξαιτία της εισαγωγή του στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση και θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για την αποψήλωση κυρίω. Εάν δείτε το χάρτη της Βραζιλίας, δυστυχώς δεν έχω έναν μαζί μου, αλλά θα δείτε ότι πρώτα απ' όλα η Βραζιλία είναι διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έκταση, σε εμπαδό. Η παραγωγή εθανόλης στη Βραζιλία προέρχεται από το ζαχαροκάλαμα, τα οποία παράγονται κυρίως στο Σάο Παόλο και στις ε, βορειοανατολικές ε, περιοχές. Η περιοχή του Αμαζονίου βρίσκεται στα βόρεια της χώρας. Η απόσταση στις περιοχές ε, μεταξύ παραγωγής εθανόλης από ζαχαροκάλαμα στη Βραζιλία και των τροπικών δασών είναι η ίδια απόσταση με την, μεταξύ Ρώμης και Μόσχας, για να σας δώσω μια ιδέα καμία σχέση δεν έχει η παραγωγή εθανόλης στη Βραζιλία με το θέμα των ε, τροπικών δασών και την αποψήλωση. Καμία σχέση. Τα μα δεν καλλιεργούνται στα δάση, αυτό είναι σαφές, ούτε σε πρώην δασικές εκτάσεις. Τώρα, για να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα, για την Τόχα. Ήδη ανέφερα ότι γύρω στη Στόκα θα περιλάμβανε μια ατζέντα με ένα κατάλογο προτεραιοτήτων με, για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων συγκεκριμένων χωρών. Τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα για τις υπηρεσίε και τι τηλεπικοινωνίε, την προστασία των εμπορικών σχέσεων και το ανέφερε ένας Ισπανός βουλευτής. Νομίζω ότι στη Βραζιλία πολλέ από τι επενδύσει στις υπηρεσίε και τηλεπικοινωνίε τηλεπικοινωνίες ε, είναι από τα σοβαρότερα μερίδια που έχουμε συνολικά στο επενδυτικό κεφάλαιο. Εάν κάνουμε μια σύγκριση στι επενδύσει, θα δούμε ότι η Βραζιλία είναι μια από τι χώρε που λαμβάνουν τι περισσότερε επενδύσει παγκοσμίω. Θέλουμε βεβαίω να συνεχίσει να αυξάνεται αυτή η τάση. Αλλά αυτό δεν μου φαίνεται παράξενο, ούτε θα παρουσιάσει ιδιαίτερε δυσκολίε. Διότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Οι επενδύσεις σε διάφορους τομείς συνεχώς αυξάνονται εδώ και κάμποσα χρόνια. Βεβαίως υπάρχουν τομείς όπου σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αυτή είναι η γραμμή που ακολουθούμε σε όλες μας τις κινήσεις ε, και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία όπω θα συνέβαινε και σε κάθε άλλη χώρα. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν εδώ σοβαρά προβλήματα ή εμπόδια. Όπου προκύπτουν προβλήματα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε αναπερίπτωση. Με επικοδομητική προσέγγιση. Τώρα τα περαιτέρω βήματα για την Τόχα. Το ανέφερα και στην ομιλία μου. εξακολουθούμε τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν προκειμένου, αλλά πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Ιδάλλως δεν έχει νόημα, δεν οδηγεί πουθενά να προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το γύρο διαπραγματεύσεων χωρίς να είναι παρόντες οι βασικοί μας εταίροι, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συζητήσεις λοιπόν, ο διάλογος εξακολουθούν. Ελπίζουμε ότι ο γύρος αυτός θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Θα ήταν καλό για το, για το εμπορικό σύστημα παγκοσμίω να γίνει κάτι τέτοιο. Για το ζήτημα της Αργεντινή και το δημόσιο χρέο. οι πληροφορίε που έχω είναι ότι άρχισαν να διαπραγματεύονται ξανά το χρέος τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, λίγο πιο σκόπιμο να το απευθύνεται ω ερώτημα στον Αργεντινό πρέσβη, σε μένα. Έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα από καιρό εις καιρόν και με αυτή την υπόθεση. Και νομίζω ότι ακόμη και στην Ευρώπη, εάν κοιτάξετε κάποιες χώρες, θα δείτε ότι είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο του χρέους, του δημόσιου χρέους και του ΑΕΠ που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Κάποιες χώρες μάλιστα έχουν περισσότερο χρέος από ότι ΑΕΠ. 100% αναλογία. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα. Η εμπιστοσύνη επιτρέπει στις κοινωνίες να περνούν στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές. Για τη βιοεθανόλη τώρα, που αναφέρθηκε από τον ίδιο βουλευτή, νομίζω το κάλυψα για τη σόγια. Υπάρχει από την Αμπιό, τη βασική μας εταιρεία, μια πρόταση συμβιβαστική. Να αποφύγουμε την αποψήλωση λόγω καλλιέργεια σόγια και να μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία αυτή είναι μια από του ένας από τους τρεις βασικούς σόγιας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ προσεκτική στην προσέγγιση του. Εγώ με ιδιαίτερη χαρά είδα πέρσι στα τέλη της χρονιάς να έχουμε τους πιο πρόσφατους αριθμούς για την αποψήλωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για την τελευταία 20 ετία τα χαμηλότερα από ό,τι ποτέ πριν. Άρα ο αγώνας που διεξάγεται κατά της αποψήλωσης δίνει καλά αποτελέσματα. Και το ερώτημα από την ε, Σουηδία. Η Σουηδία είναι σαφώς ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Βραζιλία από ευρωπαϊκής πλευράς. Αυτό μας δίνει πολλές δυνατότητες. Ξέρω ότι το Σάο Παόλο είναι από τις πόλεις που λαμβάνουν τις περισσότερες επενδύσεις από τη Σουηδία. Πολλές σουηδικές εταιρείες βρίσκονται στην ε, Βραζιλία πλέον. Κάθε φορά όμως που μιλώ για την, οικονομία της Βραζιλίας, αισθάνομαι αρκετά άνετα. Διότι έχουμε δείξει μεγάλο βαθμό ανθεκτικότητας ε, στην κρίση. Και μάλιστα περιμένουμε και μια αύξηση του, της τάξης του 5% φέτος. Τα εργαλεία λοιπόν που έχουμε προβλέψει, όπως τις ε, λήψεις, τις υποδοχής ε, επενδύσεων, δίνουν καλά αποτελέσματα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να περάσω στα γαλλικά για να πληθυνθώ στους ε, ερωτώντε ε, για την αποψήλωση και τι κλιματικέ αλλαγέ. Νομίζω ότι ήδη παρουσίασαν την τοποθέτησή μα δεν επηρεάζεται καθόλου η παραγωγή της, των ζαχαροκάλαμων από την αποψήλωση, ούτε σχετίζονται τα δύο θέματα. Τώρα, η παραγωγή εθανόλης. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται άμεσα με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό ναι, διότι ήδη αποδείξαμε με διάφορα μέσα ότι υπάρχει... υπάρχουν θετικέ επιπτώσει και εδώ μιλώ αποκλειστικά για τη Βραζιλία. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων παραγωγή που υπάρχουν ε, σε διαφορετικέ περιοχέ και για διαφορετικά προϊόντα. Στη δική μα λοιπόν ακριβώ περίπτωση, το χαροκάλαμο δεν προκαλεί, δεν απειλεί καθόλου. Δεν είναι η ίδια πρώτη ύλη άλλωστε που χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες για την παραγωγή φανόλη και είμαστε και αρκετά παραγωγικοί. Δηλαδή αν κάναμε μια σύγκριση μεταξύ της παραγωγής ε, εθανόλης από ζαχαροκάλαμο και από καλαμπόκι ε, η παραγωγή από ζαχαροκάλαμο είναι 7 φορέ πιο ε, παραγωγική από το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι ο δεν χρησιμοποιείται στην Βραζιλία και έχουμε και μια νέα μέθοδο χρήσης της καλλιεργίας αυτής για την καταπολέμηση της ρήπανσης. Για μας λοιπόν και όπως σας εξήγησα και προηγουμένως η παραγωγή όρο απέχει από τα δάση του Αμαζονίου. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τις αποστάσεις στη Βραζιλία για να το καταλάβει αυτό. Για τα γενώσιμα φάρμακα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Μία φορά αντιμετωπίσαμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με εξαγωγή φαρμάκων από την Ενδία προς την Βραζιλία. Αυτό έγινε προς τα τέλη του 2008. Και αυτό που επιθυμούμε τώρα είναι τέτοιου είδους φαινόμενα να μην επαναλαμβάνονται. Δηλαδή υπάρχουν διεθνείς κανόνες οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΠΟΗ όπως η επίσημη δήλωση τρίψ και υγεία και τα προϊόντα που αναφέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονταν σε διαμετακόμιση από την Ευρώπη. Δηλαδή πέρασαν από την Ινδία στην Ευρώπη για να φτάσουν στη Βραζιλία. Τα πράγματα αυτά είναι περίεργα. Θα πρέπει οι διεθνείς κανόνες, οι κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Τέτοιου είδους προϊόντα εφόσον είναι αντικείμενο εμπορίας, να γίνονται όλα αυτά εντός ενός πλαισίου νόμιμου. Με συγχωρείτε κύριε Πρέσβη, μπορείτε να συντομεύσετε. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο. Έχουμε μεγάλο περιορισμό. Τότε μια σύντομη μνήμα για τη σχέση της κρίσης της γης και των αποτελεσμάτων μας. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη το εξής. Όταν αναλύεται τις βραζιλιάνικες πολιτικές πώς γίνονται αντιληπτοί από τον ίδιο τον πληθυσμό της χώρας. Αυτό είναι εύκολο να το αξιολογήσει κανείς από το πώς ε, τον ε, εκτιμούν τον πρόεδρο Λούλα στην Βραζιλία. Στην ιστορία μας δεν είχαμε κανένα παράδειγμα πρόεδρου που την τελευταία χρονιά της δεύτερης θητείας του να έχει τέτοιο ποσοστό εκτίμησης από τον πληθυσμό κατά 80%. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι δείχνει ότι οι πολιτικές που έχει θεσπίσει και υλοποιεί. Και παρόλο που υπάρχει δυνατότητα βελτίωση, και υπάρχει και ένα κόστο ε, γι' αυτό, αποδεικνύει λοιπόν ότι οι πολιτικέ αυτέ έχουν δώσει καλά αποτελέσματα για τον πληθυσμό τη χώρα και για τη Βραζιλία συνολικά. Με αυτό νομίζω ότι θα κλείσω, ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και με τα χαρά, όποτε ξαναχρειαστεί, να ξαναμιλήσουμε, να ξανασυναντηθούμε για να σα δώσω περαιτέρω πληροφορίε για τα μεμονωμένα ερωτήματα που μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρέσβη. Αυτή θα είναι μόλι η αρχή μια σειρά συναντήσεων με τα μέλη τη Επιτροπής μας. Ανυπομονούμε για την επόμενη ευκαιρία. Περνάμε αμέσως στη συνάντηση των συντονιστών. Μιλάμε για μια κεκλεισμένη θηρών συνεδρίαση. Ζητώ λοιπόν από όλου όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην αίθουσα να εξέλθουν αμέσως αν γίνεται.